Η πρόεδρος κυρία Φώτιγκα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε σε μια πολύ ιδιαίτερη συνεδρίαση του σημερινού πρωινού που είναι αφιερωμένη στην αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας στα Δυτικά Βαλκάνια. Να μου επιτρέψετε όμως πρώτα να κηρύξω επίσημα την έναρξη της ε, τακτικής συνεδρίασης της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ και μετά θα προχωρήσουμε στην κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ και ΣΕΝΤΕ, δηλαδή Επιτροπής Εξωτερικών και Υποεπιτροπής Ασφαλείας. Και να σας υπενθυμίσω ότι η παρούσα συνεδρίαση, ως συνήθως, μεταδίδεται από το διαδίκτυο Παρακαλώ όμως να καθίσετε, γιατί ε, κάπως ενοχλούν οι συζητήσεις που γίνονται ακατάστατα. Σε ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώς, έχουν, έχει δοθεί προτεραιότητα στα μέλη της Υποεπιτροπής το απόγευμα για μία ώρα μεταξύ τριών και τεσσάρων ωρών θα υπάρχουν τα τσεχικά μόνο παθητικά. Ε, στην μετάφραση και λυπούμεθα πολύ γι' αυτό. Να μου επιτρέψετε τώρα να σας ζητήσω να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη για σήμερα και αύριο, για τη σημερινή και την αυριανή συνεδρία. Εάν δεν έχετε σχόλια, τότε θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Πράγματι βλέπω ότι δεν έχετε σχόλια. Και επιτρέψτε μου να σας υποβάλω τα πρακτικά της 11ης και 12ης Απριλίου. Έχετε χρόνο μέχρι τέλους της ε, συνεδρίασης της Υποεπιτροπής για να μπορέσετε να υποβάλλετε σχόλια, επιφυλάξεις και εφόσον δεν υπάρξουν σχόλια ε, θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Χωρίς άλλες ανακοινώσεις της Προέδρου, θα παραδώσω το μικρόφωνο στον κύριο Κούζο Περμόη, ο οποίος συμπροεδρεύει της ε, κοινή συνεδρίας της Επιτροπής Εξωτερικών και Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω όμως ισπανικά. Ευχαριστώ την συμπρόεδρό μου, αξιότιμη συμμετέχοντες, προσκεκλημένοι και συνάδελφοι, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την προσέλευσή σας και να σας ευχηθώ το καλώς ορίσατε στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και της Υποεπιτροπής Ασφάλειας. Θα είμαι σύντομος γιατί αυτό που ενδιαφέρει ιδίω είναι να ακούσουμε τις δικές σας σκέψεις και σχόλια. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων περνούν από μια δύσκολη περίοδο μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής και έχουν και ένα βαρύ παρελθόν. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια απειλή, διότι βρίσκονται για την ώρα σε μια ευαίσθητη και εύθραυστη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και υπάρχουν διάφορα συμφέροντα που συγκρούονται στην περιοχή τους. Πάντως σημαντικό είναι να διατηρηθεί η σταθερότητα, διότι αν δεν διατηρηθεί η σταθερότητα, οι επιπτώσεις θα είναι βαρύτατες και για την Ευρώπη στο σύνολό της, σε ό,τι αφορά ιδίω την εσωτερική ασφάλεια. Γι' αυτό και έχουμε συνέρθει σήμερα εδώ για να εξετάσουμε την κατάσταση και να δούμε τι μπορεί ενδεχομένω να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, συμπρόεδρο και να της παραδώσω αμέσως το μικρόφωνο ώστε να κάνει ε, ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συμπρόεδρε. Εξ ονόματος της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας θα ήθελα να απευθύνω τον καλό ορίσατε στους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας. Έχουμε χωρίσει το σύνολο αυτών θεμάτων σε δύο πάνελ. Στο πρώτο θα αναφερθούμε σε μια συνολική περιφερειακή επισκόπηση, την αξιολόγηση της ασφάλειας και των πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή. Το δεύτερο στοχεύει ειδικότερα σε στρατιωτικές πτυχές. Και βεβαίως το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδίως στην ασφάλεια μετά από τις στρατιωτικές παρεμβάσεις τη δεκαετίας του 1990 αναμέναμε να εξελιχθεί μια ειρηνική διαδικασία και μια σταδιακή βήμα-βήμα εξέλιξη της περιοχής με την ελπίδα να δούμε πολύ θετικά αποτελέσματα και διαδικασία Dayton και ε, βεβαίω και από τη σύνολη αντίληψη και σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς Βρισκόμαστε σε, μπροστά σε πολύ δύσκολες προκλήσεις βεβαίως και σε όλο τον κόσμο αλλά και ιδίω στα Δυτικά Βαλκάνια όπου και οι έξι χώρες που τα συναπαρτίζουν είναι, συναποτελούν μία από τις πιο περίπλοκες περιοχές της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Συχνά μιλούμε για χωνευτήρι και σίγουρα σήμερα με μια ποικιλία απειλών που βλέπουμε να εμφανίζονται όλες αυτές ξαφνικά και μάλιστα ταυτόχρονα σε πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, είτε πρόκειται για τρομοκρατικές απειλές, είτε πρόκειται για την μετανάστευση, είτε πρόκειται για την άσκηση επιρροής από την Ρωσία και τους υβριδικούς πολέμους που διεξάγει. Ιδίως λοιπόν επηρεάζουν ορισμένες από τις ε, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και η Επιτροπή Εξωτερικών και η Υποεπιτροπή Ασφαλείας μέσω των Προεδρίων τους είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν πρόσφατα με την ύπατη εκπρόσωπο καθώς και με τον Επίτροπο Χάν για την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση ασφαλείας στα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό ε, απαιτέλεσε έκκληση και προς εμάς ε, να ε, δραστηριοποιηθούμε περισσότερο. Και γι' αυτό ε, συζητούμε σήμερα μέσα στα δύο πάνελ σε κάποιο βαθμό την απάντηση που θα δώσουμε στην έκκληση αυτή και βεβαίως με παρουσία μας στην περιοχή, με πολιτικές ομάδες, με επιτροπές και με μεμονωμένους ευρωβουλευτές. Θα δώσω το λόγο τώρα πάλι στον κύριο Κούζο Περμόη για να ε, διευθύνει το πρώτο πάνελ. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το πρώτο πάνελ. Έχουμε δύο προσκεκλημένους, τον κύριο Έντουαρτ Άουερ, διευθυντή του Τμήματος Δυτικών Βαλκανίων στην Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και τον κύριο Ένταρ Φορέ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και θα παρακαλέσω τα πρόσωπα αυτά να λάβουν το λόγο με τη σειρά για 15 λεπτά και πρώτος ο κύριος Άουερ. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τις δύο επιτροπές σας για την διοργάνωση της παρούσας ε, συναντήσεως και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να μπορέσω να σας απευθύνω τον λόγο. Πριν αρχίσω να μιλώ για θέματα ασφαλείας, θα έπρεπε ίσως να πω ορισμένα πράγματα γενικά για τις σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις με τις έξι αυτές χώρες. Όλες έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική και όπως λέει και η διπλωματική μας γλώσσα, οι αρχηγοί κατών και κυβερνήσεων συζήτησαν ε, νωρίς φέτος τι σχέσεις με τα Δυτικά Βαργάνια και έχουν αναλάβει δεσμεύσει απέναντι στα Δυτικά Βαργάνια, το ίδιο και οι Υπουργοί Εξωτερικών, που έχουν και αυτοί υιοθετήσει παρόμοιε διατυπώσεις. Όλοι λοιπόν εδώ συζητούν για ασφάλεια και τις σχετικέ εξελίξεις που γίνονται στο πλαίσιο αυτών των πολύ, στενών σχέσεων με τις χώρες αυτές που έχουν, όπως είπα, μια ευρωπαϊκή προοπτική η στενότητα των σχέσεων αντανακλάται και στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, προκλήσεις παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα από τα πιο καυτά θέματα είναι οι επιστρέφοντες ε, μαχητές από Συρία και αλλού, διεθνές οργανωμένο έγκλημα, μεταναστευτικές ροές, νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και απειλές είναι η συνεργασία. Έχουμε παρόμοιες απειλές, έχουμε κοινά σύνορα με όλες τις χώρες αυτές, ώστε είναι αναγκαιότητα η συνεργασία. Και αυτό απηχείται καθαρά στην ε, σφαιρική στρατηγική που ακολουθεί στην εξωτερική πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση με στήριγμα τα, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη συνεργασία στην ε, πολιτική ασφάλειας. για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και των εξτρεμισμών. Πώς μπορεί, να πώς μπορεί να οργανωθεί η συνεργασία αυτή. Πολλά έχουν γίνει ήδη σε όλα τα θέματα που σας προανέφερα και περισσότερα από όσα θα μπορούσα να σας πω τώρα. Αλλά θα περιοριστώ σε ορισμένα από τα πιο βασικά. Ας δούμε πρώτα τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Από το 2012 έως το 2016 μεγάλος αριθμός, περίπου 950 άτομα έφυγαν από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για να μεταβούν σε Συρία και Ιράκ. Από το 2015, ωστόσο, οι αναχωρήσεις αυτές έχουν μειωθεί ε, σημαντικά. Όμως, Υπάρχουν αυτοί που επιστρέφουν σε σημαντικούς αριθμούς. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν από αυτούς που ανεχώρησαν. Ορισμένες εκατοντάδες επέστρεψαν ή μπορεί και να επιστρέψουν ακόμη και αποτελούν σημαντική απειλή. Για να αντιμετωπιστεί σωστά αυτή η απειλή, διότι πρόκειται για ανθρώπους που μπορεί να διαβούν και τα σύνορα, είναι σημαντικό οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων να μοιράζονται τις πληροφορίες που έχουν με την Ευρωπόλ, να συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο. Όλα αυτά συμβαίνουν. Χρειάζονται αποτελεσματική συνοριακή έλεγχη και ούτω καθεξής. Με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις ε, σχετικές διατάξεις στον ποινικό νόμο και στι δικαστικέ πρακτικέ. Θα πρέπει να προσθέσω ότι οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν υιοθετήσει σχετική νομοθεσία για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά. Άλλο θέμα είναι τα πυροβόλα όπλα. Από το πιο ευαίσθητο θέμα στην περιοχή αυτή, πολλά πυροβόλα όπλα έχουν παραμείνει στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μετά τους πολέμους της δεκαετίας του 90 και αποτελούν απειλή διότι είναι και εύκολη η πρόσβαση σε αυτά τα όπλα από τρομοκρατικέ ομάδε. Οι εταίροι μα των Δυτικών Βαλκανίων ε, κάνουν προσπάθειε για να αντιμετωπίσουν την, κίνηση των, ε, αυτή, την διακίνηση αυτών των πυροβόλων όπλων. Άλλο θέμα είναι τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Και εδώ χρειάζεται στενή αστυνομική συνεργασία και άλλο θέμα είναι η διαχείριση των συνόρων και ο έλεγχο των συνόρων και συνεργασία για το μεταναστευτικό. Δεν είναι πια τόσο δραστήρια η μεταναστευτική οδός των Δυτικών Βαλκανίων για τους τελευταίους 18 μήνες, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη να είμαστε ε, προετοιμασμένοι για τις εξέλιξεις. Ανέφερα ορισμένες δραστηριότητες και των ε, θεσμικών οργάνων που αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά σε συνεργασία με τις χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Θα σας δώσω μια συνολική επισκόπηση για τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει Πρώτα η Ευρωπόλ, την οποία ανέφερα, η Eurojust για θέματα ριζοσπαστικοποίησης, με ένα σημαντικό περιφερειακό πρόγραμμα το οποίο ε, διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αντιτρομοκρατική πρωτοβουλία των Δυτικών Βαλκανίων που ξεκίνησε αρχικώς από τη Σλοβενία ε, νομίζω έλεγχη για την αντιμετώπιση της διακίνησης πυροβόλων όπλων, πολύ στενή συνεργασία για τη μετανάστευση και με σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη και στο αποκορύφωμα των διαφόρων κρίσεων και τώρα διαπραγματευόμαστε συμφωνίες για τις επιχειρήσεις Frontex, ξεκινώντας από τη Σερβία. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και παρόμοιες διαπραγματεύσεις μπορεί να αρχίσουν να διεξάγονται και με άλλες χώρες. Μίλησα ήδη για το ενδιαφέρον που δείχνει το Συμβούλιο για τα Δυτικά Βαλκάνια Προ δύο ημερών, την Δευτέρα, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ενέκρινε συμπεράσματα για τις εξωτερικές αυτές δράσεις που επανεπιβεβαιώνουν την ανάγκη της ενίσχυσης της εταιρική σχέσης με τα Δυτικά Βαλκάνια για την αντιτρομοκρατία, για την αντιμετώπιση εξτρεμιστών και το παράνομο εμπόριο πυροβόλων όπλων. Επανεπιβεβαιώνουν δηλαδή στην βάση την στενή συνεργασία που έχουν οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και δίνουν τι κατευθύνσει για την περαιτέρω ενίσχυσή τη. Βεβαίω ε, βλέπουμε πρώτα τα ζητήματα ασφαλεία. Κάτι που ασφαλώς και πρέπει να έχει την προσοχή μας, αλλά χρειάζεται μια πολύ συνεκτικότερη και συνολικότερη προσέγγιση με τις ε, διαπραγματεύσεις για ένταξη των χωρών αυτών. Δύο από αυτές ε, προχωρούν ήδη. Πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες, στις οποίες εγκύπτουν οι ειδικοί οργανισμοί, αυτή η συνολική επισκόπηση είναι και η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια και σταθερότητα των χωρών αυτών, διότι τους προσφέρει ένα πολιτικό μέλλον. Προσφέρει ε, στις διάφορες πολιτικές δυνάμεις των χωρών αυτών ένα κοινό στόχο για να εργαστούν προς την επίτευξή του. Και η διαδικασία διεύρυνσης θα επιτρέψει να γίνουν και σε βάθος μεταρρυθμίσεις στις κοινωνίες αυτές. Ο κίνδυνο κατά τη σταθερότητα των χωρών της, Δυτική των, έχει μειωθεί βέβαια σημαντικά από τη δεκαετία του 1990 που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Φώτιγκα όταν οι χώρες της Βαλκανική ήταν καθημερινά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Οι απειλές έχουν μετακινηθεί τώρα προς άλλα θέματα σαν αυτά που σας προανέφερα. Έτσι, δεν φαίνονται πολύ πιθανέ νέε συγκρουσίε και κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ απίθανε και στο μέλλον και πιο μακροπρόθεσμα ακόμη. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε την επιτήρηση. Υπάρχουν στα Βαρκάνια δύο αποστολές της ΚΕΠΑ που παρακολουθούν τα θέματα αυτά στη Βοσνία Ζεγοβίνη υπό την επιχειρησιακή ε, επιτήρηση του ΝΑΤΟ και στο Κόσοβο που προσφέρει ενίσχυση στην αστυνομία, κυρίως όμως για παρακολούθηση της επιβολής του νόμου και της τάξης, ενίσχυση των δικαστικών συστημάτων κλπ. Σύντομα τώρα για τρίτες χώρες, για τη δράση τρίτων χωρών. Έχουμε σύντομη παράγραφο για το ΝΑΤΟ. Βλέπω ότι η συνάδελφος είναι εδώ και θα αναφερθεί στο θέμα για τους τις τρίτες χώρες, Ρωσία, Κίνα, Τουρκία, είναι διάφορες χώρες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με διάφορα θεματολόγια υπόψη τους. Αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης συνεδριάσεως. Νομίζω ότι υπήρξε πρώτερη ακρόαση επί των ε, τρίτων χωρών και των φορέων των τρίτων χωρών αρκεί να πούμε ότι μπορεί να υπάρξει χρήσιμη συνεργασία με κάποιους από αυτούς τους φορείς για τα θέματα των επενδύσεων, πολλές τρομοκρατίας, μετανάστευση. Πρέπει να επαγρυπνούμε όμως όσον αφορά τα προβλήματα ασφαλείας. Κάποιες δράσεις εκπροσώπων αυτών των χωρών μπορεί να δημιουργούν απειλές. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε υπερβολικά, αλλά να το έχουμε υπόψη. Για τους τρίτους φορείς, εκπροσώπους τρίτων χωρών και την πολιτική που ακολουθούν οι χώρες, Λοιπόν, κάποιε επιλέγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιε ε, το ΝΑΤΟ και πρέπει να πούμε στι τρίτε χώρε που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια ότι υποστηρίζουμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην επιλογή που έχουν κάνει. Ε, στο τέλος αναφέρω δύο θέματα. Ανέφερα κάποια θέματα επί των οποίων υπάρχει συνεργασία, κάποια πράγματα που κάνουμε. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που άφησα για το τέλος, σημαντικότατη δράση που άφησα για το τέλος. Ποια είναι αυτή? Η στατηγική επικοινωνία, μια θετική ε, διπλωματία, δημόσια ανοιχτή διπλωματία. Δεν μπορεί κανείς να την υπερεκτιμήσει. Πολλές από τις αρνητικές προπαγάνδες που προωθούνται, η αρνητική προπαγάνδα που προωθείται βγαίνει από ΜΜΕ, από ριζοσπαστικές ομάδες, και κάποιες φορές ε, από κυβερνήσεις και θα πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτό. Ευτυχώς το ποσοστό ε, ε, έγκρισης αυτών των μέτρων είναι πολύ ψηλό στα Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν υπάρχει το ακροατήριο για τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε και θα πρέπει να στείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα και να μείνουμε συνδεδεμένοι με αυτό το ακροατήριο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε να θετήσουμε στρατηγική επικοινωνία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία εξωτερική δράση έχουν εξεργαστεί για τα Δυτικά Βαλκάνια και θέλουμε να, το, να τα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα και να ενισχύσουμε ε, το κέντρο για την επικοινωνία στα Δυτικά Βαλκάνια της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως με ανθρώπους που έχουν μητρική γλώσσα των χωρών της περιοχής. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα που προσπαθούμε να προωθήσουμε. Το άλλο θέμα που ήθελα να αναφέρω στο τέλος, που είναι πολύ σημαντικό και πολύ συχνά το αγνοούμε, είναι το εξής. Παρά τις αδιαφυσβήτητες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες, καταβάλλουν προσπάθεια οι ίδιες να φροντίζουν θέματα ασφαλείας στα πλαίσια της ε, πολιτικής ασφαλείας, κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Έχουμε 15 αποστολές ε, Στατιωτικέ και πολιτικές όλο τον κόσμο και οι εταίροι μας συμβάλλουν σε νέα από αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι αρκετά αξιοσημείωτο. Εν κατακλείδη λοιπόν, να υπογραμμίσω είναι πάρα πολύ σημαντική συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ προκλήσεις μας στα πλαίσια της αφοσίωσης που δείχνει απέναντι σε αυτές τις χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κατάλληλη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα μέσα, τα υπάρχοντα δίκτυα για τη συνεργασία με τους εταίρους μας και νομίζω ότι περιέγραψα ότι ήδη διαθέτουμε πολλά εργαλεία και θα πρέπει να τα αναπτύξουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε με το σωστό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάουρ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βανφρέ, ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, μεγάλη χαρά για μένα που είμαστε εδώ σήμερα να συμβάλλω σε αυτή την ε, συζήτηση για την κατάσταση στην ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια και πραγματικά βλέποντας ε, το κλίμα αντιπαράθεσης που επικρατεί στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων είναι εύκολο να λησμονήσουμε ότι ακριβώς σε αυτή την ε, περιοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ανέπτυξε σαν ένα κομμάτι της ΣΚΕΠΑ κάποια από τα νέα εργαλεία για την ασφάλεια και την άμυνα, όπως η επιτυχής ανάπτυξη της πρώτης αστυνομικής ε, αποστολής στη Βοσνία Ζεγοβίνη το 2003 και επίσης είχαμε και την πρώτη στατιωτική επιχείρηση Κονκόρδια στο ΦΥΡΟΜ ε, τον ίδιο χρόνο. Και σε αυτή την ίδια χώρα, πριν από δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το ΝΑΤΟ και την ΟΑΣΕ κατέληξαν στη συμφωνία της Αχρίδας που έθεσε τέρμα στις συγκρούσεις της εθνοτικές στην περιοχή. Και αυτές οι εξελίξεις μαζί με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και την οικονομική υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, κατέδειξαν με ρεαλιστικό τρόπο τη δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στην ειρήνευση της περιοχής και να δημιουργήσει τις συνθήκες που επιτρέπουν στις χώρες περιοχής να προχωρήσουν προς το στόχο της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στόχο που επιβεβαιώθηκε από τη Σύνοδο Κορυφή τη Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Ενώσης το 2003. Αυτό ήταν, έγινε πριν από 14 χρόνια, πολλά συνέβησαν έκτοτε. Ε, βέβαια όλες οι χώρες της ε, περιοχής βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της ενταξιακής διαδικασίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία έγινε κράτος μέλος και ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ενταξιακές με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία και ίσως το πιο ισχυρό μήνυμα του πλησιάσματος της περιοχής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτό είναι υποφελές ε, για τους πολίτες ήταν η έγκριση Τη δυνατότητα ταξιδίων άνευ στο χώρο Σέγγεν για όλε τι χώρε τη περιοχή εκτό από το Κωσυφοπαίδιο που περιμένει ανυπόμονα να συμβεί αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε το ρόλο του στην όλη διαδικασία. Παρά αυτέ τι θετικέ εξελίξει, αναφυσβήτητα η περιοχή υπήρξε μάρτυρα στην τελευταία έτη μια σημαντική επιδείνωση όσον αφορά τι προδιαγραφέ δημοκρατικέ και αυξημένα επίπεδα διαφθορά και οργανωμένου εγκλήματο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ανακοίνωση το 2016 και αφορούσε την πολιτική διεύρυνση Ευρωπαϊκή Ενώσεω και αυτή αναφέρθηκε σε διάφορε χώρε τη περιοχή που εξακολουθούν να δείχνουν παραθέτω σαφή συμπτώματα και διάφορου βαθμού ε, παγίδευση και κρατισμού. Είτε είναι στον τομέα τη ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου, δικαιολογία των κοινοβουλευτικών θεσμών, ε, τη διαδικασία των εκλογών, τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, η επιδείνωση ήταν πραγματικά ανησυχητική και όλα αυτά έχουν καταγραφεί και έχουν καταχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΑΣΕ, την Ευρωπόλ, ε, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και άλλους διεθνείς φορείς. Και θα πρέπει να υπογραμμιστεί βέβαια ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 ε, έθεσε το κράτος δικαίου ε, στο επίκεντρο της ενταξιακής διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως η αρχή του ότι τα θεμελιώδη πρέπει να προωθούνται πρώτα, που παραθέτω λέγοντα αυτό από την τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής του περασμένου Νοεμβρίου. Αυτό ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, αλλά ακριβώς αυτούς τους τομείς βλέπουμε διολίσθηση δραματική όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Και αυτό μας εξέπληξε και αυτό οδήγησε και στην ε, δημιουργία κλίματος αντιπαράθεσης. Τα επίπεδα του οργανωμένου εγκλήματος, ε, η χρήση των ναρκωτικών, ε, το εμπόριο παράνομο των όπλων ε, είναι πραγματική πηγή ασταθείας και αυτό γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό όταν όπως είδαμε σε διάφορες ε, υποθέσεις αυτές οι δραστηριότητες προστατεύονται μέσω κρατικών και πολιτικών θεσμών. Αυτές οι εξελίξεις βεβαίως συμβαίνουν σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον ο μόνος διεθνής φορέας στην περιοχή όπως είπε και ο προλαλής σας ομιλητής ε, έχουμε αυξανόμενα επιθετική πολιτική της Ρωσίας και γίνεται αισθητή παρουσία της και στη Σερβία και στη Ρεπούμπλικα Σέρσκα. Και πέρα από τις κατηγορίες ε, ε, καζόμενης εμπλοκής σε ένα αποτυχημένο πραξικόπημα στο Μαυροβούνιο και οι προσπάθειες να τεθούν εμπόδια στην προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ για να αναφερθούμε και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Ομάδας για τη Διαμόρφωση για τα Βαλκάνια. Η κρίση της δημοκρατίας στα Δυτικά Βαλκάνια ισχύει για την αδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Τουρκία βέβαια είναι πολύ αδύναμη και χρησιμοποιεί το, την κοινή πολιτισμική προσέγγιση για να έχει επιρροή. τώρα ποιοι είναι οι λόγοι για αυτές τις αρνητικές εξελίξεις και τι δείχνει αυτό για την αποτελεσματικότητα της ε, τη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διεύρυνση προ την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Αναφεσβήτητα υπάρχουν εσωτερικέ δυσκολίε που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα, η άνοδο ε, του λαϊκισμού, τα θέματα του κατά πόσο η διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποφελή και βέβαια ε, υπήρξε και τοξική συζήτηση για τις μεταναστευτικές ροές και η ε, αποτυχία των πολιτικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να ε, προωθήσουν την επιτυχία αυτής της πολιτικής διότι φοβήθηκαν ότι θα αποξενώσουν τους ψηφοφόρους. Όλα αυτά συνέβαλαν στην αποδύναμωση τη ε, μεταμορφωτική ε, δύναμη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως και επίθεση κατά τη ελευθερία των ΜΜΕ και τη κοινωνία των πολιτών εντό τη οικογένεια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως αυτή και αυτής, όπω τα φαινόμενα που βλέπουμε στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Αυτά επίση αποδυνάμωσαν τη δυνατότητα μόχλευση και επιρροή τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως έναντι αυτών των χωρών. Η προσφυγική κρίση του 2015 με το διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών οδήγησε στην επιδίωξη συνεργασίας ε, με αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και τη σύσταση μηχανισμών μεθοριακών ελέγχων. Αυτέ οι χώρε, κυρίω η Σερβερία και η Μακεδονία, λέει ο μιλητή, βεβαίω με τα χαρά συμμορφώθηκαν, παρέχοντα μία δικαιολογία για να αποσπάσουν την προσοχή από την αυταρχική συμπεριφορά εντός των χωρών τους και ε, επιδιώκοντας αυτή την προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη εκείνα που ήταν πιο κοντά στην περιοχή δημιούργησαν την ξεκάθαρη εντύπωση ότι η εξασφάλιση σταθερότητα στην περιοχή ήταν η πρωταρχική τους μέρημνα. Το επιχείρημα τότε που προβαλόταν ήταν ότι όσο υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή, άλλε στοιχείες, όπως τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτο δικαίου ε, θα ρυθμιστούν από μόνα τους. Αλλά όπω είδαμε, στα γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία έτη, η διατήρηση σταθερότητα ει βάρο του κράτου δικαίου και της λογοδοσίας των κυβερνήσεων είναι μια συνταγή για αποτυχία μακροπρόθεσμα. Ακόμα και όταν ενεπλάκει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας ε, να ε, λύσει μια πολιτική κρίση όπως ε, στο ΦΥΡΟΜ, όταν μαζί με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξε με πολιτική συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ηγετών των κομμάτων τον Ιούλιο του 2015 δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει αποτελεσματική συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν. Αυτό παρά το γεγονός ότι μια ειδική έκθεση που ονομάστηκε έκθεση Πρίμπε και που υπευλήθη τον Ιούνιο του 2015 ε, καθόρισε σαφώς τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα για να ε, αντιμετωπιστούν συστημικές παραβιάσεις του κάτους δικαίου. Αλλά παρά την παρακολούθηση των εξελίξεων και το ότι δεν καταγγέλθησαν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αυτά τροφοδότησαν όμως το συνέστημα τιμωρησίας ε, του τότε ε, κυβερνώντος κόμματος και συνέβαλε δυστυχώς σε μία μείωση του πύχη όσον αφορά τα δημοκρατικά πρότυπα και αυτό που θεωρεί το παλιά ε, ασυνήθις συμπεριφορά θεωρήθηκε το νέο κανονικό, κανονική συμπεριφορά σήμερα. Αλλά Πρέπει να στεστούμε και στι τεχνοκρατικέ πτυχέ των μεταρρυθμίσεων, χωρί να εξετάζονται τα αίτια όμω τη διολίστηση ή το των εγκληματικών ποια ήταν η επιρροή των α, εγκληματικών δικτύων. Μην κάνοντα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την εντύπωση ότι δεν είχε μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση τη περιοχή. Αυτό επίση ε, είχε συνέπειε όσον αφορά την έλλειψη αποτελεσματική εφαρμογή των, των διαφορονομικών προδιαγραφών και των διαφόρων αναγκαίων ερευνών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και επίσης υπήρξε και μια κάποια δυναμία στην στον έλεγχο των διενέξεων. Δεν υπήρξε συστηματική υποστήριξη τη κοινωνία των πολιτών, παρά το γεγονό ότι πολύ συχνά αυτό ήταν ο μόνο φορέα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη λογοδοσία όσον αφορά του πολιτικού ηγέτε εν τη απουσία των τακτικών και κανονικών ελέγχων, που θεωρούμε κάτι δεδομένο στι δικέ μα δημοκρατικέ κοινωνίε. Αυτό επίση συνέβαλε ε, στην αδιαφάνεια και την έλλειψη λογοδοσία από πλευρά των ηγετών αυτών. Ένα διάλογο που έλαβανε χώρα κυρίω με την ελίτ πολιτική, παγιώνει την ελίτ και αγκιστρώνεται αυτή στην εξουσία παρόλο που αγνοεί τις θεμελιώδεις αξίες. Επίσης δίνει μια νομιμότητα στους ίδιους ηγέτες αυτούς. Μερικοί από αυτούς ε, τελούν υποέρευνα για εγκληματικές δραστηριότητε και κατάχρηση εξουσίας. Σχετικά με αυτό, η ύπατη εκπρόσωπος επεσκέφθη πρόσφατα τον Μάρτιο την περιοχή όπου ε, συναντήθηκε και άκουσε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και αυτό ήταν κάτι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Τώρα ποιες είναι οι λύσεις. Σας αναφέρω κάποιες από αυτές, ε, λίγες λύσεις. Το πρώτο παραθέτοντας στο Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών στην πρόσφατη διάσκεψη στο Άσπεν στο Ινστιτούτο των Υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο ορατή ε, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση από πλευρά θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και πιο συχνέ επισκέψει από του ύπατου εκπροσώπου. Ε, σχετικά με αυτό, ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιστέψει στην πρώτερη πρακτική, δηλαδή ένα επίτροπο να είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διεύρυνση και να μην έχουμε το παρόν μοντέλο συνδυάζοντα την διεύρυνση και την πολιτική γειτονία στι δύο πολιτικέ. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση θα πρέπει να μιλά πολύ πιο συχνά και πιο ηχηρά όταν οι κυβερνήσει και τα πολιτικά κόμματα αγνοούν ή παραβιάζουν ε, υποχρεώσει που έχουν αναλάβει για μεταρρυθμίσει. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στην επικοινωνία των μηνυμάτων, στην προβολή των μηνυμάτων που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να γίνεται με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, κυρίως όταν ε, αυτά μηνυματων που στελνει η ευρωπαικη ενωση και αυτο να γινεται με ανοιχτο και διαφανη τροπο κυριως οταν αυτα αναφερονται σε ε, μη συμμόρφωση με δημοκρατικές προδιαγραφές και μη μεταρρυθμίσεις πρέπει να δούμε όταν υπάρχουν παραβιάσεις στις ελευθερίες του ΜΜΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, ο εκπρόσωπος του ΑΣΕ για την ελευθερία των ΜΜΕ που είναι αυτός που εισακούεται. Ενώ πολύ συχνά ε, δεν, ηχεί, δεν αντυχεί η φωνή της Ευρωπαϊκής Ενώσης, παρά το γεγονός ότι αυτές οι χώρες είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, σε εποχές πολιτικής κρίσης που είδαμε να συμβαίνει δυστυχώς πρόσφατα, στο πρόσφατο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σοβαρά να δει ποια είναι η στρατηγική διαχείριση των συγκρούσεων, πώ να αντιμετωπίσει του πολιτικού ηγέτε που επανειλημμένα αγνοούν εκκλήσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω και που ανοιχτά δεν σέβονται τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτο δικαίου. Τέταρτον, χρειάζεται να υπάρχει αυστηρότερο έλεγχο όσον αφορά τη διαδικασία για την υιοθέτηση με ε, νομοθεσίες που αφορά μεταρρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει σωστή πρώτερη διαβούλευση με φορείς κοινωνίας των πολιτών και θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι θα παρέχονται για τους φορείς που δημιουργούνται για την εφαρμογή και υλοποίηση της νομοθεσίας. Διαφορετικά γίνεται απλώς μια άσκηση επιχάρτου όπου το Κοινοβούλιο απλώς επικυρώνει τυπικά τα μέτρα. Πέμπτον, Χρειάζεται πιο συνεπής επαφή και συνεχής επαφή με οργανώσεις της κοινωνίας των ε, πολιτών και θα πρέπει όποτε οι κυβερνήσει οι πολιτικοί ηγέτες επιτίθεται κατά αυτά των φορέων να ε, τους επικρίνουμε και όταν επίσης δέχονται επιθέσεις. Η επαφή με την κοινωνία των πολιτών ε, εξασφαλίζει πιο ληστική προσέγγιση στον αφορά τη συζήτηση Ευρωπαϊκή Ένωση με την περιοχή. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό σε εποχέ μια κρίση ένα θετικό παράδειγμα σχετικά με αυτό είναι το σχέδιο για κατεπίγουσες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που υθετήθηκε πέρσι εν το μέσο της μακεδονικής πολιτικής κρίσης νομιλητής με πάνω από 70 οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που ήταν κάτι επρόσδεκτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεση χωρών του Νοεμβρίου. Έκτον, θα πρέπει να υπάρχει πιο ενεργή προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση διμερών διαφορών, ιδιαίτερω εκείνων που εμπλέκουν ξεχωριστά Όσον αυτές οι διαφορές παραμένουν ανεπίλητες, τόσο πιο πολύ υπονομεύουν την αξιοπιστία της ε, διαδικασίας διευρύνσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κυρίως το, το στοιχείο της δικαιοσύνης όσον αφορά την αρχή της αρεσιμότητας. Επίσης, τροφοδοτεί την το εθνικιστικό θεματολόγιο των ε, χωρών των Βαλκανίων που συζητούμε. Έβδομον, χρειάζεται να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες αντιμετώπιση των απαραδεκτών υψηλών επιπέδων ανεργία των νέων, κυρίως που φτάνει 60% σε κάποιες χώρες. Με χωρί, αν δεν υπάρχουν προπτικές για απασχόληση, αποξενώνεται η νεολαία, κυρίως σε κάποιες χώρες όπως το Κωσυφοπέδιο και η Βοσνία Ζεγοβίνη, που γίνονται στόχος ε, για ε, να τους ε, στρατολογήσουν οι ξένοι μαχητές για τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας και άλλη μια πηγή σταθείας. Όγδον η διαδικασία του Βερολίνου, που είναι πρόσδεκτη η πρωτοβουλία της Γερμανίδας Καγκελαρίου του 2014, έδωσε ε, ιδιαίτερη προσοχή στην περιφερειακή ε, συνεργασία, κυρίως στη ασυνδημότητα, όσον αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές, συμπεριλαμβάνοντας τις πανευρωπαϊκούς διαδρόμους. Τα θέματα που αφορούν το κάτω δικαίου και δημοκρατική διακυβέρνηση θα πρέπει περισσότερο να προωθούνται από τούδε στο εξή στα επόμενα στάδια της διαδικασίας και κυρίως στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Τεργέστη. Αν δεν υπάρχουν κράτος δικαίου, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο και θα ωφελήσουν μόνο τους λίγους και θα αφήσουν έξω τους πιο ευάλωτους και κυρίως την νεολαία. Κάτι που είδαμε την ανεργία. Και όπως ο ίδιος είπε ο Επίτροπος Χαν στο επιχειρηματικό φόρουμ τον περασμένο Ιούλιο, το κράτος δικαίου και οι οικονομικές εξελίξεις είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Πιστεύω ότι ένα αποτελεσματικό τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις πολλές αδυναμίε που παρουσιάστηκαν θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα συμμετάσχει μέσω ελέγχου ή μέσω πραγματικών διαπραγματεύσεων ε, σε μια διαδικασία με όλες τις χώρες της περιοχής στις περιοχές που καλύπτονται από τα κεφάλαια 23 και 24 τη διαδικασία ένταξη. Και αυτό θα κρατήσει σε μια αλληλεπίδραση τι χώρε που έχουν κάνει αίτηση με του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, εφόσον είμαστε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερε προσπάθειε από τι μεγάλε πολιτικέ οικογένειε που είναι παρούσε εδώ για να δημιουργηθεί μια πιο όρημη πολιτική κουλτούρα και σεβασμό για τα δημοκρατικά πρότυπα στα αδελφά κόμματα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και να επιβάλλονται κυρώσει σε αυτού που παραβιάζουν αυτά τα πρότυπα ή που οι ηγέτες τους ε, είναι αντικείμενο ποινικών ε, ε, ερευνών. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κλείνοντας να πω και δύο λόγια ελπίδας στην στρατηγική για την ε, στη συνολική στρατηγική για την ΚΕΠΑ της, ε, είπα, της εκπροσώπου πέρυσι δηλώνεται ότι ε, μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επένδυση για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης και πάντοτε συνεισέφερε στην ειρήνη σε περιοχές που είχαν στο παρελθόν μαστίζονταν από πόλεμο. Άρα εστιάζοντας περισσότερο στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τελευταίες εβδομάδες, όχι μόνο ε, στις σημερινές συνεδρίες αλλά και γενικότερα, αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας, δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, για τις ε, επικίνδυνες τάσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Μια περιοχή που έχει παραγάγει μεγάλα κομμάτια ιστορία περισσότερο από όσα μπορεί να απορροφήσει. Και μόνο αποκαθιστώντα την αξιοπιστία στην πολιτική διεύρυνση και με μια πιο συνολική στρατηγική λύση θα μπορέσει να καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απομακρύνει τα φαντάσματα των Βαλκανίων του παρελθόντο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ας αρχίσουμε την συζήτηση. Μπορείτε να μου ζητήσετε τον λόγο εφόσον θέλετε να παρέμβετε. Ο κύριος Πέτερλε είναι ο πρώτος ε, ομιλητής εκ των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα δύο μέλη του πάνελ για τις ε, σαφείς τοποθετήσεις τους. Συμφωνώ ότι μιλούμε για μια περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας και βεβαίως στρατηγικές περιοχές χρειάζονται και στρατηγική συμπεριφορά και στρατηγικές πολιτικές κατά κάποιο τρόπο. Κατέστησα σαφές τα τελευταία χρόνια ότι δεν μπορούμε να ενισχύσουμε αξιόπιστα την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων εάν φανούμε αδύναμοι στον πυρήνα, εάν οι Βρυξέλλες είναι αδύναμες. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ελπίζω ότι μετά τις εκλογές θα, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ξανά την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι ο κινητήρας, ο γαλλογερμανικός κινητήρας θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, να αρχίσει πάλι να αποδίδει. Εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία του Βερολίνου που αναφέρατε πριν, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι ένα καλό εργαλείο για να προωθηθεί η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών. Όσο δεν βλέπουν παρουσία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης οι χώρες αυτές, τόσο θα καλύψουν το κενό άλλοι παίκτες εντό εισαγωγικών. Ε, είναι ώρα λοιπόν να γίνουν επενδύσεις, να επενδυθούν πολιτικά. Νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η διάσταση ασφαλείας. Πριν από 20-25 χρόνια μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ επενδύσαμε πολύ στην σταθερότητα για να πάυσουν οι πόλεμοι, ιδίως στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να γίνουν προσπάθειες για το λεγόμενο nation building, για να σταθούν αυτά κράτη στα πόδια τους. Είναι σημαντικό να υπερβούμε δύο ασυμμετρικές καταστάσεις ή μάλλον πολύ ασυμμετρικές καταστάσεις όπου ορισμένες χώρες κάνουν κάποια πρόοδο, άλλες μένουν πίσω, αλλά όλες ανήκουν στην ίδια περιοχή. Και με την εξαίρεση της Αλβανίας ανήκαν πριν στην ίδια χώρα. Πρέπει να βρούμε τρόπους λοιπόν, εκεί όπου δεν κατέστη δυνατή πρόοδος έως τώρα, πρέπει να αναζητήσουμε άλλε στρατηγικέ για να διευκολύνουμε την πρόοδο. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, αλλά έχουν τόσο διαφορετικά καθεστώτα οι υποψήφιε χώρε, αφού το Κόσοβο ούτε καν είναι υποψήφια χώρα, δεν μπορούμε να πετύχουμε πολύ πρόοδο. Και νομίζω ότι πρέπει να προσφέρουμε μια καλύτερη δυναμική και όπως είπε ο κύριος Φουερέ στα τελευταία 7 σημεία του, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρόσφατα ηγήθηκα στο Κόσοβο αντιπροσωπείας για την παρατήρηση των εκλογών και είδα πόσο έντονο είναι το παρελθόν ακόμη στην περιοχή αυτή. Μόνο εάν μπορέσουμε να εμπλέξουμε φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στην περιοχή αυτή με καθαρή στατική και καθαρή πολιτική. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτελέσουμε πρόοδο. Αλλιώς θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αργότερα. Θυμούμε πώς ήταν τα πράγματα πριν από 26 χρόνια στη δική μου χώρα, τη Σλοβενία. Είχαμε πόλεμο που μετά μετα, μετακινήθηκε στην Κροατία και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να ξαναδώ τέτοια πράγματα στην περιοχή μας. γνώρισα, δεν θέλω να κάνω χιούμορ σήμερα, αλλά τέλος πάντων ε, εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, αλλά γνώρισα κάποιον που μου είπε Αλόης, πρώτα Brexit και μετά Δυτικά Βαλκάνια. Εμένα δεν μου αρέσει έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι ευγνώμων στους δύο μιλητές που έλαβαν το λόγο μας έδωσαν μία ακριβή εικόνα και ευχαριστώ ιδίω τον πρέσβη Φουερέ για την ιδιαίτερα επακριβή και λεπτομερή αξιολόγηση που μας έκανε. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι στην περιφέρεια, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι ρίζες. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο κύρια προβλήματα. Πρώτον, το status quo. Την Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχεθήκαμε τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια και δεν τα καταφέραμε να κάνουμε μια αληθινή διαδικασία διεύρυνσης, να είναι μια απτή διαδικασία που θα δίνει προοπτική ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες αυτές και τώρα έχει προαπαινθεί στις ελληνικές καλένδες. δεν μας αρέσει είτε όχι, δεν υπάρχει κάποια προοπτική πλέον. Δεύτερον, υπάρχει μια νέα διαδικασία ε, στους ε, λαούς της περιοχής η επικράτηση της ε, σταθερότητας. Νομίζουν οι πολίτες ότι αν μείνουν οι ηγέτες για μεγαλύτερο χρόνο στην εξουσία θα επικρατήσει σταθερότητα. Αλλά αν δεν υπάρχει και επαρκές κράτος δικαίου και σωστή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, δεν είναι θετικό το να παραμένουν οι ηγέτες στην εξουσία. Μπορεί να είναι και αρνητικό, να είναι παράγον κινδύνου. Αν δείτε τις εξελίξεις σε ορισμένες περιοχές όπου επενδύσαμε στη διατήρηση της σταθερότητας, δημιουργούνται κίνδυνοι. δεν αποκομίζουμε ωφέλη. Αντιθέτως, πρέπει να ε, καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για τη σταθερότητα στις περιοχές αυτές. Επίσης υπάρχει και μια κόποση, μια κόποση στην πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένε χώρες, αλλά για τις περιοχές αυτής της περιφέρειας υπάρχει μια τοξική κόποση. Η κόποση του ότι έχουν αναμείνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολλούς λαούς της περιφέρειας η διαδικασία διεύρυνσης δεν φαίνεται να είναι απτή και πραγματική. και όσον αφορά την πολιτική διάσταση και όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα με την οποία η διαδικασία διεύρυνσης ε, έχει επιπτώσει στην πραγματική καθημερινή ζωή των ανθρώπων στην περιφέρεια. Σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε. Και δέχομαι ότι εμείς τα πολιτικά κόμματα στο Κοινοβούλιο έχουμε τις ευθύνες μας και φέρουμε κάποια ευθύνη για την περιφέρεια αυτή. Αντί να υποστηρίζουμε ανεφόρον τα πολιτικά μας κόμματα στην περιφέρεια αυτή, θεωρούμε ότι οι δικοί μας ηθήνοντες είναι καλύτεροι από τους δικούς τους ηθήνοντες και όσο δεν εκφέρουμε κριτική και δεν υποστηρίζουμε ε, τα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα, διακινδυνεύουμε να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική ένταση και ακόμη περισσότερο ε, αντιφατικές πολιτικές όπως ε, περιστατικά βίας στην Μακεδονία λέει ο ή στην Βοσνία ή στην Σερβία. Ε, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες ε, δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν έχει σημασία αν κάποιος ηγέτης είναι σοσιαλιστής αλλά ε, είναι κοντά στην πολιτική ομάδα του ΕΛΚ. Αν κάποιοι ηγέτες δεν είναι επαρκείς δεν θα πρέπει να τους υποστηρίζουμε και η δική μας συμπεριφορά, η συμπεριφορά των δικών μας πολιτικών ομάδων φέρει κάποια ευθύνη για την κατάσταση στην περιφέρεια. Και τέλος δεν θα πρέπει απλώς να αρκούμεθα στα μεγάλα λόγια αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να δημιουργηθεί ένα επαρκές οικονομικό πακέτο μέτρων για μια οικονομική αναδιάρθρωση της περιοχής με αυτοκινητοδρόμους, ε, με ενεργειακές οδούς για να υπάρξει μεγαλύτερη ολοκλήρωση στην ευρωπαϊκή αγορά. Διότι αυτό είναι και το πρωταρχικό στοιχείο μιας πραγματικής διαδικασίας διεύρυνσης. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει το θεματολόγιο της διεύρυνσης να το προωθήσουμε και να μην ε, το αφήνουμε να γίνεται όμοιρος της εθνικής πολιτικής όπως γίνεται στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, η διαδικασία χάνεται, η διαδικασία διεύρυνσης γίνεται όλο και πιο αδύναμη και οι υπόλοιποι φορείς, η Ρωσία, Κίνα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, θα κερδίσουν τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σκέλα Σκέλαμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ χρήσιμη και επίκαιρη αυτή η ανταλλαγή απόψεων, διότι οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι έχουμε κοινέ ανησυχίες και κοινά συμφέροντα. Τα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι μόνα τους. Έχουμε προγράμματα και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθερότητα της περιοχής. Καλά προγράμματα που προσφέρουν ασφάλεια. Αλλά είναι σαφές σήμερα, όπως είπε και ο κύριος Μποστινάρο προηγουμένως, ότι σημειώνεται κόποση και από την πλευρά της Ένωσης και κόποση και απογοήτευση από την πλευρά των χωρών που έχουν υποβάλει αιτήσεις ένταξης. Το βασικό είναι ότι οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση να συνεχίζεται όπως είναι, διότι είναι ένας φαύλος κύκλος χωρίς καθαρή προοπτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε διστακτική, καμιά φορά αμφίθυμη. Δεν μπορούμε ούτε να συνεχίσουμε σαν να είμαστε δάσκαλοι και μαθητές να κάνεις τα μαθήματά σου γιατί αλλιώς, α, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Διότι αυτά τα βήματα αποτυγχάνουν και είναι η κοινή μας ευθύνη να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές. Εγώ υποστηρίζω πολύ την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια ισχυρότερη και πιο ορατή παρουσία. Μιλήσατε για ειδικό επίτροπο που να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο με ειδικό αντικείμενο αυτή την περιφέρεια. Δεύτερο, το ερώτημα πώς αντιμετωπίζουμε τις ξένες επιρροές. Ρώσος απεσταλμένος στην ε, Μακεδονία, σύμφωνα με τον ομιλητή, τελευταία, λέει ότι θέλει να προσφέρει νέα προοπτική στις χώρες αυτές. Σωστά είπατε ότι η Ρωσία δεν έχει ισχυρή οικονομία. Έχει όμως. Παίζει τα δύναμα χαρτιά της με τρόπο δυνατό, εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άλλα μέρη που ενδιαφέρονται. Ρωσία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε ένα καθαρό πρόγραμμα. Και επανέρχομαι στον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφασιστικότητα για να συμβάλλει στη ρύθμιση των θεμάτων. Μετά για διμερείς εθνικές συγκρούσεις. Το 2001 η Μακεδονία βρισκόταν στα πρόθυρα ένοπλης σύραξης με Αλβανία. Πώς μπορούμε να δείξουμε το δρόμο εδώ, διαμεσολαβώντας στις ε, αντιπαρθέσεις αυτές. Και τέλος, αυτή η μετακομμουνιστική περιοχή, που έχει όμως ολόκληρο το παρελθόν πολύ σημαντική επιρροή στην οικονομική διαφθορά, με ισχυρές ομάδες πώς μπορεί ε, να προωθηθεί μια συμφιλίωση της περιοχής με το παρελθόν. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να δοθεί. Διότι αλλιώς συχνά αυτή η ατζέντα, το, θεματολόγιο της ελεύθερης αγοράς για τον τόπιο πληθυσμό τους φαίνεται πιο πολύ να είναι η ατζέντα των καινούριων μαφιόζων και των ε, ομάδων εξουσίας που παίζουν τα παιχνίδια τους εκεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Και υποστηρίζω ένθερμα τα επλογηθέντα σχόλια του κυρίου Μποστινάρου και το τελευταίο που είπε ο κύριος Κίλαμ. Αυτό που με εξέπληξε από την παρουσιάση σα ήταν αυτό που είπε ο κ. Άιλ για τις θετικές επαφές με το λαό, με το κοινό και να ενισχύσουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας στην περιφέρεια. Ακούγοντας αυτά που είπε ο κ. Φιέ, βλέπουμε ότι το θέμα αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Τις αξίες που προβάλλουμε και κατά πόσο εκπροσωπούμε δημοσία τη σημασία και το βάθος των αξιών. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας που προβάλλουμε μέσω της επικοινωνίας. Άρα, η ερώτησή μου θα ήταν εκεί, η εξής. Ποια είναι η ανταπόκριση σας στη σχόλια του κυρίου Φίρερ. Για το πώς μπορούμε να κινηθούμε πιο ενεργά και πώς μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα στα μηνύματα που προβάλλουμε. Υπογραμμίζοντας πάντα τις αξίες μας. Η επικοινωνία και η στρατηγική να βασίζεται στις αξίες μας. Αυτό είναι το βασικό. Ευχαριστώ κύριο Σκούκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευπρόσδεκτη συζήτηση. Συζητούμε στην Επιτροπή μας πολλά σημαντικά θέματα. Το θέμα της ασφαλείας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι περιπλοκότατο ζήτημα. Ευχαριστώ και καλωσορίζω τους συγκεκριμένου καλεσμένους μας και ευχαριστώ πολύ για την κατάσταση που τον τρόπο παρουσίασαν την κατάσταση. Είναι επίκαιρη συζήτηση, όπως είπε ο συνάδελφος ΛΑΜ την περασμένη εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο συζήτησε τα προβλήματα και τα ζητήματα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Τα θέματα ασφαλείας της περιοχής πρέπει να τα προσέξουμε περισσότερο είναι πολύ συνδεδεμένη με την περιοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν περιφέρεια, αλλά να απόσπαστο κομμάτι της δομής που έχουμε για την ασφάλεια. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε και τα θέματα ασφαλείας, προλήψεως συγκρούσεων και ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου. Ασφάλεια δεν αφορά μόνο μόνο τη διαχείριση απειλών και συγκρούσεων, αλλά να έχουμε παρόμοια προσέγγιση για θέματα ασφαλείας. Πολύ συχνά ακούω ανησυχίε σχετικά με αυτό, όσον αφορά ε, τις εθνοτικές εντάσεις, όπως τη Μακεδονία, Λεωμιλητής, Κωσυφοπαίδιο, Βοσνία, Ζεγοβίνη και πώς ε, κινείται το οργανωμένο έγκλημα και τι γίνεται με το εμπόριο όπλων. Στα πλαίσια της ενταξιακής πορείας των χωρών μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς την εξωτερική πολιτική και την αντιμετώπιση ασφαλείας, να ευθυγραμμιστεί η κίνηση και η θέση αυτών των χωρών με τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει να τα προωθήσουμε αυτά πιο ενεργά. Άλλη ανησυχία. Η επιρροή άλλων διεθνών παικτών στην περιφέρεια. Σε κάποιες χώρες βλέπουμε ισχυρή παρουσία της Ρωσίας, σε άλλες χώρες ισχυρή παρουσία της Τουρκίας. πρέπει να κινηθούν προς συλλογική άμυνα και ασφάλεια αυτές οι χώρες. Ολόκληρη η Αδριατική ακτή της Αδριατικής ανήκει στο ΝΑΤΟ και ελπίζω η Μακεδονία, λέει ο σύντομα να γίνει μέλος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι τα λέμε αυτά επί πολλά χρόνια. Λέγαμε ότι περιμένουμε σύντομα να προχωρήσουν οι χώρες. Θα ήταν καλό λοιπόν αυτό πραγματικά να γίνει σχετικά με αυτό. Επανειλημμένα θα πρέπει να στέλνουμε ισχυρά πολιτικά μηνύματα προς τους εταίρους της περιοχής. Να τους λέμε ότι οι προσανατολισμοί τους για ασφάλεια και εξωτερική πολιτική πρέπει να στρέφεται προς τις Βρυξέλλες. Εκτιμώ τις εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις των δύο δικαιωμένων καλεσμένων μας. Άκουσα με μέγιστη προσοχή τις δέκα εντολές ούτως υπήν του κυρίου Φουερέ, του κυρίου Πρέσβη. Μου άρεσαν αυτά τα σημεία, εμπεριείχαν ευφιέστατες ιδέες. Κύριε Πρέσβη, με τα λύπης μου λέω ότι δεν θα εφαρμοστούν αμέσως όλες. Αν είστε ρεαλιστής θα το κατανοείτε. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις ιδέες που αναφέρατε. Πολλές φορές συζητώντα τα Δυτικά Βαλκάνια. Τέλος. Εκτιμούμε και κατανοούμε την κατάσταση, κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η περιοχή και προτείνουμε πολλά θετικά για να βοηθήσουμε όμως πρέπει να θυμόμαστε πάντα ποια είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Βάγκελ. Ah. Έχει ερώτηση. Θέλει, θέλετε να μιλήσετε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Πρώτα, το θέμα της ευθύνης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι ευθύνες κάποιων χωρών μελών σχετικά με την ασφάλεια των Δυτικών Βαλκανίων, της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε φτάνει καθυστερημένη απέναντι στις εξελίξεις στην περιοχή αυτή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ή το ΝΑΤΟ μας προλαβαίνει πάντα. Έτσι έγινε και στον πόλεμο των Βαρκανιών. Χρειάστηκε η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. για να οδηγήσει σε λύση. Είχαμε και πάλι την εμπειρία ότι και τώρα το ΝΑΤΟ είναι πριν από μας παρόν, δέχεται την συμμετοχή ως πλήρους μέλους του Μαυροβουνίου και στο πόσο από πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν προλάβει. Έχουμε τεράστια ευθύνη κάτω από αυτές τις περιστάσεις ασφαλείας. Για παράδειγμα, οι πέντε χώρες που δεν αναγνώρισαν το Κόσοβο έχουν, φέρουν ευθύνη για την κατάσταση. Ή η Ελλάδα στην περίπτωση της Μακεδονίας κατά τον ομιλητή. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στην δημιουργία, στην πρόκληση της μακεδονικής κρίσης, εμείς είμαστε οι πρώτοι υπεύθυνοι, εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αναβάλουμε διαρκώς την ένταξη της Μακεδονίας και η Ελλάς μπλοκάρει την ένταξη της Μακεδονίας. Εμείς λοιπόν καλούμεθα να κάνουμε περισσότερα. Η δική μας συνεισφορά είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της περιοχής. Ευχαριστώ κύριε Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι οι προλαλήσαντες ε, ανέλησαν πολύ παραστατικά και με ακρίβεια τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα Δυτικά Βαλκάνια. Ιδιαίτερα επισημαίνω και συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο Μποστινάρου, ο οποίο όχι μόνο επισήμανε τα προβλήματα, αλλά έδωσε και λύσει πρακτικέ, οι οποίε μπορεί να γίνουν σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να αρχίσουν. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και να διαφωνήσω σαφώ με την τοποθέτηση του τελευταίου συναδέλφου σχετικά με το γιατί τα Σκόπια δεν γίνονται ακόμη αποδεκτά στην Ευρώπη και για το γεγονός βεβαίως ότι ευθύνη φέρουν και για τις υπόλοιπες πέντε χώρες, εκείνες οι χώρες οι οποίες δεν τις έχουν αναγνωρίσει. Ας αρχίσουμε από το τελευταίο. Οι πέντε χώρες οι οποίες δεν αναγνωρίζουν αυτές τις χώρες οι οποίες θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το Κόσοβο, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα, δεν το κάνουν ούτε για λόγους αντιδράσεως, ούτε διότι δεν υπάρχει λόγος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Κωσυφοπαίδιο αυτή τη στιγμή αποτελεί μία από τις πλέον διεφθαρμένες χώρες της, Ευρωπα... της Ευρώπης και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και να αναγνωριστεί από κάποιες χώρες οι οποίες έχουν το λόγο τους το κάνουν αυτό το πράγμα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα Σκόπια. Τα Σκόπια πέραν του ότι προσβάλλουν την Ελλάδα με το να χρησιμοποιούν το ιστορικό όνομα της χώρας, το ξέρετε όλοι, εκφράζουν και επεκτατικέ βλέψει κατά τη Ελλάδο. Πώ είναι δυνατόν λοιπόν η Ελλάδα να αποδεχθεί τέτοια πράγματα. Αν ήταν η χώρα η δική σα ή η χώρα του κυρίου συναδέλφου, αυτή η οποία υφίστατο αυτή την πρόκληση, θα αντιδρούσε διαφορετικά. Θα δεχότανε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και στο ΝΑΤΟ, μια χώρα η οποία θα έχει δικαίωμα βέτο όταν αυτή η χώρα διεκδικεί εδάφη τη δική σου χώρα. Από την άλλη πλευρά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο απέναντι στις χώρες οι οποίες παραβιάζουν σαφώς και τη, δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και εν πάση περιπτώσει δεν έχουν κατορθώσει να δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση ώστε να έχουν τη δυνατότητα και να πληρούν τα κριτήρια για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι αντιμετωπίζουμε τις χώρες αυτές με τέτοια φιλοσοφία να κάνουμε κάτι τίποτε διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνει κάποιος ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσει ενός κακομαθημένου παιδιού πιστεύοντας ότι αυτό στο τέλος θα κάνει εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει. Με τέτοια νοοτροπία δεν πρόκειται να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα Δυτικά Βαλκάνια διότι πάνω απ' όλα δεν θα υπάρχει ομοφωνία και συνένεση από τις χώρε οι οποίες θίγονται από την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά. Ευχαριστώ. Ο Συμπρόεδρος, μία παρατήρηση πιο πολύ για την ασφάλεια ωστόσο. Έχουμε, μάλλον ακούσαμε, ότι 950 μαχητές απεχώρησαν από τις χώρες αυτές για να μεταβούν στη Συρία και στο Ιράκ να πολεμήσουν εκεί. Πόσοι επέστρεψαν και πόσοι κινήθηκαν προς τις περιοχές του Καυκάσου. Αυτό θα ήθελα να μου απαντηθεί αν είναι δυνατόν. Και τι γίνεται με τη συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η συνεργασία με την Ρωσία. Κάποιος εκ των ε, ομιλητών αναφέρθηκε στο Κόσοβο. Νομίζω ότι έχουμε όντως διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις. Υπάρχει όμως ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και θα συνεχίσουμε να το τηρούμε. Θεωρώ ότι αυτά προκαλούν πολλά προβλήματα και είμαι πεπισμένος ότι η μόνη λύση μπορεί να βασίζεται στο διάλογο Ε, κυρία Φωτιγιά. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα δύο μέλη του πάνελ, τους δύο προσκεκλημένους, για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις τους, διαφορετικές στο χαρακτήρα του κυρίου Άουερ, κάπως πιο ήπια σε τόνο, ε, αφού παρουσιάζει κάπως την ματιά των θεσμών, σύντομη και νομίζω προσεκτικά διατυπωμένη του κυρίου Φουερέ θα έλεγα ότι ήταν ε, πραγματικά θαυμάσια διατυπωμένη με πολιτικό χαρακτήρα αλλά και με έμπνευση και επειδή με ε, Πολωνέζα διαφωνώ, διαφωνώ με τη δήλωσή σας περί Πολωνίας αλλά θα διατηρήσω την θέση μου και θα συνεχίσω να προεδρεύω χωρίς να εμπλακώ στη συζήτηση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε, ιδίω εν ώψη και της επικείμενης Βρετανικής αποχώρησης και της πολύ σημαντικής εμπλοκής των Βρετανών στα Δυτικά Βαργάνια, χρειαζόμαστε μια θετική ισορροπία στην ασφάλεια, στην οποία συνέβαλε η Βρετανία. Χρειαζόμαστε πολύ προσεκτική αξιολόγηση των θέσεών μας. Πρέπει να μην δυσμονούμε πόσο ευαίσθητη είναι η κατάσταση ασφαλείας εκεί, πόσο πολλές είναι οι προκλήσεις, πόσο πολλά είναι τα σημαντικά θέματα που παίζουν ρόλο και θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζουμε Βεβαίως και πολλά σφάλματα δικά μας. Να προσπαθήσουμε κατά κάποιο τρόπο να δώσουμε αφετηρία σε θετικές διαδικασίες και εξελίξεις σε όλη την περιοχή. Πρέπει δηλαδή να αναζητήσουμε τις θετικές πλευρές. Όμως οφείλουμε να γνωρίσουμε επίσης ότι ήταν τεράστιο σφάλμα από την αρχή ήδη της θητείας να πούμε όχι περαιτέρω διεύρυνση στο προβλεπόμενο μέλλον. Βεβαίως όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό εννοεί και τα Δυτικά Βαλκάνια και ε, υπέστη με ε, σημαντική κριτική και από άλλες χώρες ε, από τα Ανατολικά, Ουκρανία για παράδειγμα και νομίζω ότι αυτό οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασης για τη διαδικασία της, για τις χώρες μάλλον της διαδικασίας της Και ένα άλλο πράγμα θα πρέπει εξετάζοντας τη συνολική κατάσταση της περιοχής να δούμε βέβαια τις θετικές διαδικασίες προσπαθώντας να μην συμβάλλουμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η τελική έγκριση της ένταξης ε, στο ΝΑΤΟ του Μαυροβουνίου ήταν πάρα πολύ θετική. Και οι άλλοι εταίροι του ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι η εμπλοκή στην Αλβανία είναι πάρα πολύ θετική και πολύ θετική εξέλιξη. Δεν θα πρέπει ωστόσο να λησμονούμε την ασφάλεια, ιδίω την άμυνα και τη στρατιωτική εμπλοκή χωρών όπως η Σερβία. Και όταν προσπαθούμε να φέρουμε κοντύτερα τις χώρες αυτές, πρέπει να τονίζουμε αυτά που περιλαμβάνονται και στην έκθεση, θαυμάσια έκθεση για την Σερβία του David McAllister, και για την κριτική που ασκήσαμε στις πρόσφατες ασκήσεις που έκανε η Σερβία με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, που η Λευκορωσία είναι κοντά στα πολωνικά σύνορα. Και βεβαίως τα υβριδικά συνθήματα της Ρωσίας που όταν θέλει να ασκήσει επιρροή στην Ουκρανία και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη μιλούν, οι Ρώσοι, για τη σλοβενική πίστη των χωρών αυτών. Και αυτές οι ασκήσεις που έγιναν και κατά των σλαβικών εθνών στην πραγματικότητα, με τα συνθήματα αυτά. Καθαρά υβριδική δράση δηλαδή, και οφείλουμε να το έχουμε υπόψη αυτό. Και ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, βγήκε και επέκρινε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Συμπρόεδρος. Ας ακούσουμε τους ε, ε, δύο δύο να απαντήσουν με ανάποδη σειρά τώρα για πέντε λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν το λόγο και σχολίασαν. Εκτιμώ τα μάλα τα σχολιά τους. Δεν θα σχολιάσω τα πάντα. Θα επιληφθεί κάποιον σημείο ο συνάδελφος. Ένα-δύο σημεία να θίξω. Κάποιοι ομιλητές τόνισαν το εύθραυστον των θεσμών στα Δυτικά Βαλκάνια. Όλοι συμφωνούμε. Και το ιστορικό βάρος. Αυτή η περιοχή σίγουρα έχει περισσότερο ιστορικό βάρος από, τις, από πολλές περιοχές στον κόσμο και εξακολουθεί να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις σήμερα. Και όπως αναφέρθηκε και στο Κωσυφοπέδιο σε κάθε γωνιά του δρόμου υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Βλέποντας την ιστορία της Ευρώπης, εκεί σε κάθε σελίδα σχεδόν αναφέρονται τα τελευταία 100 χρόνια τα Δυτικά Βαλκάνια. Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των προγραμμάτων υποστήριξης, κυρίως για την κοινωνία των πολιτών, για την οικοδόμηση των κρατικών δομών, ό,τι σχετίζεται με τη δασκαλία της ιστορίας. Αν δείτε τα βιβλία ιστορίας σε κάποιες από τις χώρες αυτές, προωθούν μυσαλλοδοξία, μίσος, ε, προωθούν ε, διάφορες ε, διχαστικές προσεγγίσεις. Επαναλαμβάνουν κατά κάποιο τρόπο την ιστορία. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ σοβαρό, κυρίως για τις νεότερες γενιές. Υπάρχει ένα έξοχο πρόγραμμα, το Κέντρο της Θεσσαλονίκη για τη Δημοκρατία, που προωθεί ιστορικά βιβλία, διδασκαλία της ιστορίας και κοινά ιστορικά βιβλία για την περιοχή. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία που θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο, διότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Να βοηθήσει πια ανοιχτή προσέγγιση όσον αφορά την παιδεία στις χώρες της περιοχής. Αντίστοιχη με την ανάγκη εξυγχρονισμού και αντιμετώπιση του παρελθόντος και εξοικείωση με το παρελθόν. Και αυτή η εξοικείωση και συμφωλίωση με το παρελθόν είναι κάτι που είναι δυσχερέστατο. Σε πολλές κοινωνίες μετά από συγκρούσεις και στη χώρα μου, στην Ιρλανδία, πρέπει να περάσουμε από διαδικασία συμφιλίωσης. Αλλά είναι δυνατόν, είχα το προνόμιο να είμαι μάρτυρας της διαδικασίας συμφιλίωσης σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και στη Νότια Αφρική και υπάρχουν ένα-δύο έξοχα προγράμματα συμφιλιώσεως που προωθούνται τώρα από κοινωνία των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, Ρίκον, η πρωτοβουλία Ρίκον το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τέτοια πρωτοβουλία είναι καλή. Συμφιλίωση είναι επιτυχής μόνο αν έχει ρίζες στην περιοχή. Δεν μπορεί να επιβληθεί, όμως είναι μια κρίσιμη πτυχή που πρέπει να προωθηθεί για την ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει να υπάρξει συμφιλίωση με το παρελθόν, να επουλωθούν οι πληγές του παρελθόντος, αλλά να αναπτυχθεί και ένα αφήγημα το οποίο μπορεί να στερνηθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να μην επαναλαμβάνει το μίσος, να ξεπερνά το παρελθόν, να προωθείται ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Θα περιοριστώ σε αυτά στα σχόλιά μου, ελπίζοντας το ευχολόγιο μου οι δέκα εντολές. Όπως είπε ο κ. Κούκαν, κάποιες από τις εντολές μου τουλάχιστον θα καρποφορήσουν και ίσως θα εμπνεύσουν τους λαμβάνοντες αποφάσεις να σκεφτούν τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως συντομότατα αναφέρω τρία σημεία. Κάποιες ερωτήσεις εθέθησαν αφορούσαν πόσο αφοσιωμένε είναι στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Αν φαίνεται απόμακρη ενταξιακή διαδικασία. Οι εταίροι μας στα Δυτικά Βαλκάνια εκφράζουν παρόμοιες ανησυχίες με αυτές που εξεφράσαν εδώ. Τι να πω. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το σκοπό. Έχουμε ε, μία πολιτική και στατική διεύρυνση. Προχωρούμε σταθερά. Προωθούμε όλε τι δημιουργούμε θεσμού. Προωθούμε μεταρρυθμίσει όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τα προωθούμε αυτά στι διαπραγματεύσει, τα στοιχεία. Υπάρχει η προσέγγιση, υφίσταται η πολιτική μας, την προωθούμε. Άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα έθεσαν οι ομιλητές. Διαφορά μεταξύ σταθερότητος και κράτους δικαίου. Αν στηρίζουμε το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχει επιλογή μεταξύ των δύο. Όσον αφορά το κράτος δικαίου. Ε, με το κράτος δικαίου κοινωνία εγγυάται μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζεται από αυτό. Κάποιος ανέφερε το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΦΥΡΟΜ τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Προσπαθήσαμε να συναθρήσουμε τις, τα πολιτικά κόμματα να αποδεχτούν κοινούς κανόνες και να πάνε προς εκλογές σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και να συμφωνήσουν με σημαντικό πακέτο μεταρρυθμίσεων Τεράστια προσπάθεια κατεβλήθη για τη στήριξη του κράτους δικαίου, από βράση θεωρητικής τουλάχιστον, και μεταρρυθμίσεως των θεσμών. Κανείς δεν ήξερε τα αποτελέσματα των εκλογών, πολλούς εξέπληξαν τα αποτελέσματα, ότι η πρώην αντιπολίτευση νίκησε. Εσιαστήκαμε κατά πολύ σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθηθεί η δημοκρατική διαδικασία. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα των προσπαθειών. Οι γειτονικέ χώρε, η Αλβανία, τα δύο-τρία τελευταία χρόνια καταβάλουμε έντονες προσπάθειες για μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, του συστήματος δικαιοσύνης, κάτι που υιοθετήθηκε σαν νομοσχέδιο πρόσφατα από το Κοινοβούλιο, σκληρή διαδικασία, ξοδέψαμε πολύ χρόνο αλλά αν το πετύχαμε θα αλλάξει ο δικαστικός κλάδος, θα αλλάξει το προσωπικό, οι δικαστές, οι εισαγγελείς. Και αυτό είναι ένα μήνυμα πολύ σαφές για τη στήριξη του κράτους δικαίου. Τέτοια πράγματα πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμη σταθερότητα, για την επικοινωνία. Η κυρία Μούντι είπε ότι πρέπει να εξετάσουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ακριβώς. Αυτό ξετάζουμε τα μηνύματα είναι ελκυστικά για τους πολίτες. Έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά αποδοχή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και έγκριση Ευρωπαϊκή Ενώσεω στην περιοχή. Άρα τα περισσότερα μηνύματά μα είναι σωστά, φαίνεται. Πιστεύουμε ότι ακολουθούμε σωστό δρόμο. Τι πρέπει να προσέξουμε. Κάτι που Αυτά που προβληματίζουν άμεσα τους πολίτες. Να τους δείξουμε το πώς η ολοκληρώση οδηγεί σε περισσότερες ελευθερίες για τα ταξίδια, κράτος δικαίου, καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτά είναι τα θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους πολίτες των χωρών. Και αυτό πρέπει να προβληθεί σαφώς στα μηνύματά μας. Όχι αφηρημένα, με συγκεκριμένου όρους να καταλάβει ο κόσμος. Και γι' αυτό Μιλάω και για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Είναι σημαντικό το στοιχείο των προσπαθειών επικοινωνίας. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Οπότε ολοκληρώσαμε τη συζήτηση και δίνω το λόγο στην συνάδελφο για το επόμενο πάνελ. Ας χειροκροτήσουμε τους ομιλητές μας. Like to thank both. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συμμετέχοντες στη συζήτηση και θα ήθελα τώρα να καλέσω τρεις διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους μας για το δεύτερο τμήμα που αφορά ε, την ε, κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Πριν σας παρουσιάσω τους επόμενους ομιλητές, θα ήθελα να πω δύο λόγια διαδικαστικά ε, θέλω να καλωσορίσω την Κλέρ Μούντι σε αυτή τη συνάντηση, την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και θέλω να σας ενημερώσω ότι η κυρία Μούντι ορίστηκε από την ομάδα των σοσιαλιστών ε, ως αντικαταστάτρια του κυρίου Αυσαν Καν, ε, αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, ΣΕΝΤΕ που εξελέγει πρόσφατα στην ε, <clears throat> Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο. Ε, καλωσορίζουμε λοιπόν την καινούργια ε, Ευρωβουλευτή μας και θα συνεχίσουμε με τη διαδικασία εκλογών τον Ιούλιο. Ξέρουμε ότι η κυρία Μούντι έχει οριστεί για τη θέση του Αντιπροέδρου. Ευχαριστώ πολύ.

for Ladies and gentlemen, please. Καθίστε κυρίες και κύριοι και πάλι. Και περνάμε στο επίσης πολύ ενδιαφέρον δεύτερο τμήμα αυτής ε, της ε, ανταλλαγής απόψεων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε στενή συνεργασία με την Επιτροπή ΑΦΕΤ και με τον Συμπρόεδρο κ. Κούσο Περμόη και σε αυτό το δεύτερο τμήμα θα ήθελα να παρουσιάσω τους δύο συμμετέχοντες. Θα έρθει και ε, ο τρίτος συμμετέχον, οπότε θα τους παρουσιάσω και τους τρεις. Έχουμε τον στρατηγό Sir James Everard, που είναι αναπληρωτής, είπα, το συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και όπως έλεγα και σήμερα το πρωί, για πρώτη φορά έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον υποστράτηγο Τζοβάνι Φούγκο, διοικητή της δύναμης για το κοσυφοπαίδιο του ΝΑΤΟ. Έχουμε λοιπόν ε, προσκεκλημένους πολύ υψηλού επίπεδου και ε, τρίτη συμμετέχουσα, ο πρέσβης Δραγκάνα Ραντούλοβιτς, επικεφαλής της αποστολής του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ. Μόνιμη εκπρόσωπος του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ ήδη. που θα μας ενημερώσει, ελπίζω όχι μόνο για την κατάσταση στο Μαυροβούνιο, αλλά εν μέρη και για τη διαδικασία διαπραγματεύσεων, διότι ήταν επικεφαλής της ομάδας διαπραγματεύσεων του Μαυροβουνίου για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Την καλωσορίζουμε λοιπόν και χωρίς ε, να καθυστερήσουμε περαιτέρω, εδώ έχουμε συγκεκριμένες αξιολογήσεις για συγκεκριμένες χώρες, άρα οι διακεκριμένοι ομιλητές μας θα παρουσιάσουν την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα θέματα της επιλογής τους. Δίνω τον λόγο στο στρατηγό Everett και στη συνέχεια υποστράτηγο Giovanni Φούγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διακεκριμένη Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, είμαι εδώ ω ε, διοικητή των επιχειρήσεων τη ε, U4 της ε, επιχείρηση Althea. Έχω μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μου για μια σύντομη ενημέρωση για την τωρινή κατάσταση στη Βοσνία Ρεζεγοβίνη και για την επιχείρηση Althea που υποστηρίζεται, όπω γνωρίζετε, με τη χρήση κοινών στοιχείων ενεργητικού και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ και θα σας ενημερώσω και για την ε, συμμετοχή μας ε, στην ε, στρατηγική επισκόπηση που γίνεται υπό την Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού. Θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι διότι από το 1995 υπό τα Ηνωμένα Έθνη έχει επιβληθεί και διατηρηθεί με επιτυχία η ειρήνη και σιγά σιγά μειώνονται οι αριθμοί των ε, στρατευμάτων που απασχολούμε, μειώνεται το κόστος και η κατάσταση ασφάλειας ε, βελτιώνεται συνεχώς καθώς βελτιώνονται και οι ικανότητες των εθνικών ε, αρχών επιβολής της τάξης. Η EU4 είναι σχετικά φθηνή επιχείρηση, αλλά είναι μια απαραίτητη επένδυση και στην πράξη και ψυχολογικά για την υποστήριξη των αρχών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος και για να έχουμε μια καλή εικόνα της περιοχής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα η EU4 θα μπορούσε ε, με βάση τις συστάσεις της στρατηγικής επισκόπησης να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ε, συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο ε, εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέσβης Βαγγεμάρκ, έχει πει ότι το μέλλον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στο απόμακρο μέλλον, αλλά μέσα στη δική μας γενιά και έτσι και πρέπει να γίνει αν θέλουμε να αλλάξουμε την ε, κατάσταση το ότι η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι η χώρα με τα υψηλότερα επίπεδα μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα όπου η υποστήριξη του λαού για ε, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ισχυρή. Δεν είναι κάτι που θα γίνει μέσα σε μια νύχτα γιατί υπάρχουν βαθιά ριζωμένα προβλήματα στην κοινωνία αλλά δεν υπάρχει και άλλη εναλλακτική λύση και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά τα δικά μας μηνύματα για την ανάγκη για μεταρρύθμιση με βάση τις αρχές της αιρεσιμότητας για να ενημερώσουμε, να ενθαρρύνουμε και να εμπνεύσουμε αναγνωρίζοντας ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ισχυρότερο όσο περισσότερο οι πολίτες πιστεύουν ε, στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι βέβαια εύκολο. Η σταθερότητα και η πρόοδος στη Βοσνία Ζεγοβίνη παραμένει σημαντική, Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον Ντέιτον και εγώ ήμουν επικεφαλή ταξιαρχία το 1995 στη Βοσνία Ζεγοβίνη και θυμάμαι ότι ο πρέσβη Χόλμπρουκ περιέγραφε τον Ντέιτον ε, σαν μια ε, απαραίτητη ε, δομή, ένα κατασκεύασμα το οποίο ήταν αποτέλεσμα αναγκαιότητας. Εκτότε ε, είχαμε πολιτικό διέξοδο στη Βοσνία Ζεγοβίνη και με πολλές ε, εκλογικές διαδικασίες υπάρχει στασιμότητα. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική συμφιλίωση και ε, η αιστεία στο παρελθόν είναι καταστροφική. Είναι πολύ ευάλωτο η ισορροπία μεταξύ των εθνοτικών ομάδων και οι πολιτικέ ελίτ φαίνεται ότι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμβιβασμό και ενδιαφέρονται περισσότερο σε σημειακέ νίκε μεταξύ του. Επίση, στη μεταρρύθμιση βλέπουν κάποιο κίνδυνο για τη δική του εξουσία και το δικό του γόητρο. Δεν είναι πολυσυλλεκτικέ ή ε, προοδευτικέ και το πολιτικό πελατειακό κράτο ε, είναι έντονο. Τα αποτελέσματα του οργανωμένου εγκλήματο στη διαφθοράς του εξτρεμισμού και των εξωτερικών, ε, αρνητικών εξωτερικών ε, επιδράσεων είναι επίση αρνητικά, όπω και τα μέσα ενημέρωση που έχουν εθνοτικέ και πολιτικέ κατευθύνσει. Αν δεν υπάρξει λοιπόν πολυσυλλεκτική ηγετική τάση, το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα υπάρχουν πολλέ αντιπαραθέσει και όχι πολιτική συνεργασία δεν υπάρχουν κάποιοι άμεσοι κίνδυνοι, αλλά θα μπορούσε να επανέλθει μια κατάσταση ε, εθνοτικών διενέξεων. Η αποστολή, ε, η αποστολή μας, ε, η επιχείρηση Άλθια, καλύπτει πολλά στοιχεία, αποτροπή καθώς και συμμόρφωση για να πληρούμε το ρόλο ο οποίο ορίζεται στι συμφωνίε του Ντέιτον και του Παρισιού για την υποστήριξη τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να διατηρήσει ένα ασφαλέ και προστατευμένο περιβάλλον, παρέχοντα παράλληλα δυνατότητε ε, ενίσχυση δυναμικού και εκπαίδευση τη ε, ένοπλε δυνάμει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Υπάρχουν έξι βασικοί στόχοι, όπως βλέπετε στην ε, διαφάνεια που προβάλλεται. Και παρότι οι στόχοι αυτοί αφορούν ε, τις ε, επιχειρήσεις εντός του θεάτρου επιχειρήσεων, έχουν και στρατηγικές επιπτώσεις. Εκτός από τις εφαιρετικές δυνάμεις, έχουμε περίπου 550 στρατιώτες ε, επιτόπου. Είναι πολύ μικρή ε, η δύναμη U4. Ε, το 43% είναι στο MNBN και μία από τις υπομονάδες αφορά την προστασία των δυνάμεων. Είναι πολύ περιορισμένες λοιπόν οι δυνάμεις που έχουμε. Και παρότι το μέγεθος είναι μικρό, η παρουσία της EU4 και αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω έχει δυσανάλογα μεγάλο, δυσανάλογα θετικό αποτέλεσμα για τον ε, πληθυσμό επιτόπου και για τη διεθνή κοινότητα. Γνωρίζουν ότι η EU4 είναι το άκρο του δόρατος είναι μια σχέση με στρατιωτικές δυνάμεις ισχυρότερες εάν απαιτηθεί. Και αυτή ε, είναι η δύναμή της, γιατί το αποτέλεσμα είναι να εξασφαλίσει τους πολλούς και να αποτρέψει τους λίγους σε μια εποχή που αυτό συνεισφέρει άμεσα στο να διατηρηθεί το ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Αυτό είναι όλο και περισσότερο σημαντικό, διότι η συνεργασία με τις διοπτικέ αρχές βελτιώνεται μεν, παρόλα αυτά παραμένουν εμπόδια από τις διαφορετικές ερμηνείε του νόμου και από τις πολιτικές ε, παρεμβάσει. Θα γνωρίζετε επίσης ε, ότι έχουμε και εφεδρικέ δυνάμεις σε ετοιμότητα. Υπάρχει κάποια, ε, κάποιο έλλειμμα στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς μόνο ένα τάγμα είναι διαθέσιμο από τα τρία τα οποία ε, υποτίθεται ότι υπάρχουν στο σχέδιο της επιχείρησης που έχει εγκριθεί. Αυτό αποτελεί μια δυναμία και θα συνεχίσω να ζητώ από όλες τις χώρες να καλύψουν αυτό το έλλειμμα και ίσως με βάση τα αποτελέσματα της στρατηγικής επισκόπησης να εξετάσουν μια ευρύτερη ε, δυνατότητα ε, ενίσχυσης στην περιοχή. Ε, θα ήθελα να μιλήσω επίσης και για την ε, ετοιμότητα. Οι ασκήσεις ε, και οι επιχειρησιακές ασκήσεις και τα σχέδια δείχνουν ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ετοιμότητά μας και να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας. Η άσκηση Quick Resolve του 2016 έδειξε ότι έχουμε καλά αποτελέσματα. Η ικανότητά μας να χρησιμοποιήσουμε τις εφεδρικέ αυτές δυνάμεις βασίζεται στην σωστή εικόνα που έχουμε για την κατάσταση επιτόπου. Η u 4 εξέτασε την κατάσταση πρόσφατα και έχουμε κάνει αρκετές βελτιώσεις, ιδίως ε, για το Κέντρο Κοινών Επιχειρήσεων και για τις 17 ε, ομάδες συνδέσμου και παρατήρησης. οι ομάδες αυτές ε, συνδέσμου και επιτήρησης ε, μας παρέχουν αυτό που θεωρούμε βασικές πληροφορίες. Ο στρατηγός Άντων Βάλτνερ, διοικητής των δυνάμεων, καθώς και εγώ πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνολική μας προσέγγιση ώστε να έχουμε μια συνολική ε, εικόνα, μια συνολική αντίληψη, επεκτείνοντας το δίκτυό μας και βελτιώνοντας ε, το σύνδεσμό μας με το ΝΑΤΟ, με τις ε, αρχές επιβολής του νόμου επιτόπου, με τις περιφερειακές οργανώσεις ασφάλειας και με τη διεθνή κοινότητα. Η υπεροχή ανάπτυξης ικανοτήτων και εκπαίδευσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την U4. Ε, Έχω ζητήσει να γίνει επακριβής ε, υπολογισμό του αποτελέσματο, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο δεδομένων όλων των φορέων που εμπλέκονται, που είναι οι ένοπλε δυνάμει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και διεθνεί ε, φορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και υπάρχει δυσκολία στο συντονισμό των προσπαθειών εκπαίδευσης ε, που διεξάγεται. Έχουν συμμετάσχει όμως ε, το 75% των αξιωματικών των ενόχλων δυνάμεων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης σε κάποια προγράμματα κατάρτισης ε, και έχουμε εκπαιδεύσει και αρκετούς εξειδικευμένους έχουν συμμετάσχει ε, και στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, στο Κονγκό και στο Μάλι και στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Απαιτείται η πλήρης υλοποίηση ε, της επισκόπησης άμυνας και συνεχής συνεργασία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο και αν υπάρχει ένα ενιαίο σημείο από το οποίο θα γίνεται ο συντονισμός, τα αποτελέσματα θα είναι πιο καλά. Όσον αφορά ε, τα ε, κριτικά και τον εξοπλισμό, η U4 συνεχίζει την επιτήρηση και επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν μονάδες ελέγχου στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Το 2016 η U4 υποστήριξε ε, την άρση πάνω από 2.500 ε, τόνων πυρομαχικών, 96% του στόχου, αλλά παραμένουν ε, μεγάλες ποσότητες αποθηκευμένες και παραμένει ε, το έργο εν εξελίξη είναι πολύ καλό το γενικότερο σχέδιο παρόλα αυτά. Όσον αφορά την άρση των ναρκοπαιδίων, η U4 θεωρεί ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει τα μέσα ε, να επιτύχει την άρση των ναρκών και μηχανισμών, αλλά δεν έχει την απαραίτητη βούληση για να το κάνει. Μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο και να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η Βοσνία Ζεγοβίνη ε, πιστεί σε αυτό το καθήκον. Όσον αφορά τη στρατηγική επισκόπηση, συμφωνούμε με την Διεύθυνση διαχείριση Κρίσεων και Σχεδιασμού και ο πολιτικός σύμβουλος της U4 εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και υποστηρίζει την Διεύθυνση διαχείριση Κρίσεων και Σχεδιασμού για το έργο αυτό. Έχουμε υποστηρίξει την ε, επίσκεψη ε, στο Σεράγεβο ε, από πλευράς της CMPD και έχουμε ολοκληρώσει το έργο της συλλογής πληροφοριών για να εξετάσουμε το επίπεδο εκπλήρωσης της εντολής της επιχείρησης Άλθια τα, οι διαπιστώσει μα είναι ότι υπάρχει πολιτικό διέξοδο και υπάρχει στασιμότητα στην πρόοδο στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Δεν υπάρχει πιθανότητα άμεση ε, διένεξη μεταξύ των εθνοτήτων, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό μετανάστευση ε, και δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο μέλλον. Παραμένει υποστήριξη ε, για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η U4 είναι σχετικά μη δαπανήριο αλλά απαραίτητο μέσο και θα πρέπει η U4 να προσαρμοστεί με βάση τα αποτελέσματα και τις συστάσεις που θα υποβληθούν από τη στρατηγική επισκόπηση, ούτως ώστε να ενισχυθεί η συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη στρατηγική επισκόπηση που θα μας δώσει τη σωστή λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, στρατηγέ και παρακαλώ δεχτείτε τη συγγνώμη μας διότι σας διαθέσαμε λίγο χρόνο. Ε, αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος σας ε, στα διαδραματιζόμενα στη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, είναι μεγάλη τιμή για μένα που έχω τη δυνατότητα να απευθύνω το λόγο σε τέτοιο διακεκριμένο ακροατήριο για ένα τόσο ε, σημαντικό και ευαίσθητο θέμα όπως είναι η ασφάλεια του Κωσόβου. Δέκα μήνες ε, τώρα είμαι διοικητής της Κόσοβο Φως, της δύναμης που είχε ε, ιδρυθεί το 1999. Θα σας πω πού βρισκόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα από άποψη ασφαλείας. Πρώτα, όταν μιλώ για Κόσοβο, το εννοώ ως περιοχή επιχειρήσεων αρμοδιότητας της K4 σύμφωνα με το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Φάιρομ εννοώ πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και οι απόψει μου είναι απόψει της K4 και όχι απαραίτητα επίσημες απόψεις του ΝΑΤΟ. Ποια είναι η K4? είναι η μακροβιότερη επιχείρηση του ΝΑΤΟ έως τώρα, έχοντας ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 1999. Βλέπετε κάποιες πρόσφατες εικόνες τώρα ε, από τις δραστηριότητες των ανδρών και γυναικών της K4 σε όλο το Κόσοβο που δρούν και επιχειρούν υπό παντός είδους ε, συνθήκες και με μηδενικές και κάτω από το μηδέν θερμοκρασίες, χιόνια κλπ. Ποια είναι η K4? Η K4 είναι διεθνής δύναμη με σημαντική συμμετοχή του ΝΑΤΟ. Η μακροβιότερη επιχείρηση του ΝΑΤΟ έως τώρα και πλέον επιτυχής αρχίζει με 55.000 στρατιώτες το 1999, έχει κατέβει τώρα στις 4.500 στρατιωτικούς. Αποτελείται από 29 χώρες, 20 από αυτές είναι και μέλη του ΝΑΤΟ Εννέα δεν είναι. Και η περισσότερη δύναμη προσφέρεται από χώρες που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια, ένα ειδικό μείγμα κινητικών και μη κινητικών ικανοτήτων και τι εννοώ, κινητικές εννοώ διαρθρωμένη κλασικά στρατιωτική δύναμη που είναι σε θέση να κάνει όλες τις θετικέ δραστηριότητες και μη κινητική, non-kinetic, είναι μικρές μονάδες οι οποίες ζουν κοντά, πολύ κοντά στις τοπικές αρχές του Κωσόβου και παρακολουθούν το τι συμβαίνει στην κοινωνία του Κωσόβου. Άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η K4 ιδρύθηκε αρχικά για να καθιδρύσει, να διατηρήσει και τώρα να συμβάλλει σε περιβάλλον ασφαλείας στο Κόσοβο και σε ελευθερία κινήσεων, freedom of movement. Και γι' αυτό μεταφέρεται τώρα η ευθύνη στις τοπικές αρχές του Κόσοβου για την ε, ίδια ασφάλεια. Είμαστε πρώτη, τρίτη security responder, δηλαδή αυτοί που ανταποκρίνονται σε κρίσεις ασφαλείας, μετά την KP και την ULEX. Η KP είναι η πρώτη που αντιδρούν για την ίδια την ασφάλεια του Κωσόβου. Εάν δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τότε ζητούν παρέμβαση της EULEX. Εάν η EULEX ούτε αυτή είναι ικανή να αντιμετωπίσει, τότε ζητούν παρέμβαση της K4. Είναι σαφές για όλους στην περιοχή ότι αν η K4 αναπτύξει στρατιωτικό προσωπικό σε επιχείρηση για να στηρίξει KP και EULEX, στους δρόμους της Πρίστινα σε άλλες πόλεις του Κωσόβου σημαίνει ότι σημαίνει οπισθοδρόμηση. Αυτό πρέπει να τονιστεί διότι συχνά η μη ανάληψη δράσης αποτελεί επιτυχία. Στηρίζουμε και την ανάπτυξη του Κοσόβου και ΕΣΟ για την, για την δημιουργία τοπικών ικανοτήτων, local capacity, και τη διεθνή κοινότητα. Οργανισμούς αντιμετώπισης επιγουσών καταστάσεων, ό,τι μπορεί να συμβεί στο Κόσοβο δηλαδή, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της Kosovo Security Force μέσα στα όρια της δικής τους εντολής. Δηλαδή πρόκειται για δύναμη οργανωμένη για να παρέχει προστασία πολιτών και καθήκοντα προστασίας πολιτών στηρίζουμε και την διεθνή κοινότητα. Έχουμε θαυμάσια σχέση ιδίω με την EULEX, που είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των προσπαθειών του ΝΑΤΟ και των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση της ασφάλειας, για την εγγύηση μάλλον ασφάλεια του Κωσόβου. Η αποστολή της ΚΕΙΦΟΡ. Στη βάση της είναι το ψήφισμα 44 των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται τώρα για πολιτική στασιμότητα που δεν έχει επιτρέψει να εφαρμοστεί πλήρως πρακτικά το 1244, το οποίο παραμένει αμετάβλητο από το 1999. Όλα τα σχετικά έγγραφα λοιπόν ξεκινούν από το 1999, καθώς και η Τεχνική Συμφωνία για τη βελτίωση των σχέσεων με την K4 και με τις Serbian Security Forces παρακαλείται ο μιλητή να διαβάζει λίγο αργότερα. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά αρχικά και δεν προλαβαίνουμε να τον παρακολουθήσουμε. Αν είναι δυνατόν να το επισημάνει κάποιο. Θεωρείται λοιπόν η αφετηρία της μετατροπής των Κόσοβο Security Forces στη μελλοντική, στο μελλοντικό στρατό του Κόσοβου. Τώρα, εμβαθύνουμε στον ρόλο και στα καθήκοντα της K4 που συνεχίζει να δρά σαν ουδέτερος εγγυητής της σταθερότητας με ειδικό καθεστώς απέναντι στους θεσμούς του Κωσόβου και από την άποψη αυτή η K4 θεωρείται από τους Αλβανούς του Κωσόβου σαν εγγυητής κατά των απειλών και εγγυητής κατά εσωτερικών απειλών. Και σύμφωνα με το 1244 των Ηνωμένων Εθνών η K4 ελέγχει και τα σύνορα τα διοικητικά σύνορα που θεωρούνται πραγματικά σύνορα τώρα από την πλευρά του Κωσόβου και διοικητικά σύνορα μονάχα από την πλευρά της Σερβίας. Κάνουμε συγχρονισμένες περιπολίες με τις σερβικές στρατιωτικές δυνάμεις και με την ε, αστυνομία του Κωσόβου. Σύγχρονα patrols, δηλαδή υπάρχει μια περιπολία της K4 η οποία βαδίζει μαζί με τις περιπόλους των Σέρβων και με στοιχεία της K4 και της αστυνομίας του Κωσόβου που διεξάγουν ταυτόχρονα αστυνομικές επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε κάποια προβλήματα, διότι συχνά η παρουσία μας δεν γίνεται δεκτή από τις σερβικές στρατιωτικές δυνάμεις. Διότι αν δεχθούν την πολύ εγγύης παρουσία στο σύνορο, σημαίνει ότι αναγνωρίζουν την κυριαρχία της περιοχής. Η K4 παρέχει ασφάλεια στην Μητρόβιτσα και στην Πρίστινα με στόχο να μεταφερθούν τα καθήκοντα αυτά στις αρχές του Κωσόβου. Ήδη όμως από το 1999, για να κάνω μια σύγκριση, και η ΦΟΡ φύλαγε 150 static sites, ενώ τώρα αυτές έχουν μειωθεί σε αριθμό. Εν τέλει, υπάρχει και τακτικό εφεδρικό τάγμα της K4 έτοιμο να δραστηριοποιηθεί σε περίπτωση που το ζητήσει η EU4. Έγινε και συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα. Το K4 εξασφαλίζει την ασφάλεια όχι μόνο μέσα στο Κόσοβο, αλλά ακτινοβολεί σταθερότητα και σε όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Σύντομη λοιπόν επισκόπηση αυτή ήταν του ότι κάνει το ΚΕΙΦΟΡ. Τώρα ας έρθουμε στην κατάσταση ασφαλείας στο Κόσοβο. Ασφάλεια στο Κόσοβο δεν μπορεί να θεωρηθεί σε απομόνωση. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη και οι υπόλοιπε συνθήκε ασφαλείας στην όλη περιοχή. Το Κόσοβο και τα Δυτικά Βαλκάνια αντιμετωπίζουν πολλέ πηγέ αστάθεια. Η ΚΕΙΦΟΡ τι αντιμετωπίζει αυτέ σε καθημερινή βάση. Πρώτα, πολιτικές και διεθνωτικές εντάσεις, όπου ο λόγος πολλών πολιτικών τρέφει τις εντάσεις αυτές μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων και διεξάγεται πραγματικός πόλεμος συμβόλων. Πόλεμος χωρίς όπλα, αλλά με σύμβολα. Που εξαρτάται πολύ από την σημασία που το αποδίδουν τα μίδια με εντάσεις μεταξύ Πρίστινα και Βελιγραδίου και εννοώ ότι υπάρχουν συμβολικά σημάδια του περιβάλλοντος στο ε, Κόσοβο τα οποία προάγονται από τα μίδια για να εμπλέκουν τη διεθνή κοινότητα στις εξελίξεις μεγαλύτερο ρόλο παίζει ο τοπικός εξτρεμισμός. Από το Κόσοβο και μόνο 3.400 αλλοδαπή μαχητές. Φτώχεια, ανεργία, κοινωνία με αποκλεισμούς και παρόλο που οι θεσμοί στο Κόσοβο έχουν εγκρίνει νομοθεσία για την πρόληψη, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα πράγματα και κυρίως όσον αφορά ε, αποτελεσματικά προγράμματα απορριζοσπαστικοποίησης θα δούμε τους, πρώτους, ε, τους επόμενους μήνες τους πρώτους αλλοδαπούς μαχητές να αρχίσουν να απολύονται από τις φυλακές έχοντας εκτίσει τις ποινές τους και να επανέρχονται στην κοινωνία. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Επιρροή από τη Ρωσία στην περιοχή. Δεν επηρεάζει άμεσα κανένα κίνημα, έχει έμεση προσέγγιση με ισχυρή ρητορική υπέρ σλαβικών κινημάτων και με διάδοση fake news. Μετανάστες. Το Κόσοβο δεν είναι κατά μήκο της ε, Βαλκανικής οδού. Μέχρι τώρα το Κόσοβο λοιπόν λίγους ε, παράνομους μετανάστες έχει δει που κυρίως περνούν μέσα από το Κόσοβο πηγαίνοντας προς τη Σερβία και μετά προσπαθούν να φτάσουν στη Βόρεια Ευρώπη. Οι μετανάστες στο Κόσοβο ωστόσο μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα εφόσον εγκαταστούν σε περιοχές που δεν έχουμε ακόμα πλήρη έλεγχο. Εν τέλει, τα εγκλήματα πολέμου. Πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Με βαθιές εντάσεις μεταξύ των ε, κοινοτήτων. Ασφάλεια των μαρτύρων στις ε, δίκες του Διεθνούς Δικαστηρίου Οι πρώτες διώξεις πρόκειται να αρχίσουν ήδη φέτος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση ασφαλείας στο Κόσοβο σε έναν φαύλο κύκλο. Πολιτική αστάθεια φάνηκε και από τις πρόσφατες εκλογές. Παρεμοδίζουν το διάλογο μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου βίος εξτρεμισμός το Βελιγράδι αμφισβητεί αλλά και μέρη των κοινοτήτων του Κόσοβου τη μετατροπή του ΚΕΣΕΦ στη μελετικό στρατό του Κόσοβου και αυτά οδηγούν σε σημαντική αστάθεια και στο Κόσοβο και στην ευρύτερη περιοχή είναι έφραυστη και ασταθής η κατάσταση και είναι δυνατόν να κλιμακωθεί ταχύτατα η βία. Εμπλοκή και της Γιούλεξ, ε, ξαναλέω ότι εδώ είναι ουσιώδης εταίρος της k και οι προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας και αυτοί όλοι είναι σημαντικοί παράγοντες για την ασφάλεια του Κόσοβου. σημαντικό εργαλείο είναι η προσέγγιση με τον ΝΑΤΟ για την διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή. Πολλές προκλήσεις αντιμετωπίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με το Κόσοβο και πρώτα η K4 προσπαθεί να διατηρήσει την πρόσβαση με τις βόρειες κοινότητες του Κόσοβου που είναι σχεδόν ε, μονολυθικοί πληθυσμοί από Σέρβους του Κόσοβου Πρόκειται για τέσσερις κοινότητες. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αποδοχή από τον KSF και ιδίως για τα καθήκοντα εκείνα που είναι ουσιώδη για τις τοπικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, ε, αφοπλισμός ναρκών, ε, έρευνα και διάσωση. Ο διάλογος δεν είναι ακόμα επιτυχής. Στόχος είναι η πλήρης ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου, μεταξύ Σέρβων και υπολείπων Κωσοβάρων. Στο ίδιο επίπεδο που εντείνονται οι σχέσεις μπορεί να υπάρξουν και αρνητικές εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διατηρήσει τον διάλογο και η ΚΕΙΦΟΡ την στηρίζει. Η παρουσία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεν είναι απλά απλοτακτικό θέμα συνεργασίας μεταξύ K4 και EULEX, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά κατά πολύ αυτά και μπαίνει στο πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς εξακολουθούν να βρίσκονται στη βάση των περισσότερων προβλημάτων δύο συγκρουόμενες θέσεις. Πλήρης ανεξαρτησία όπως λέει η Πρίστινα, ή εδαφική ακαιρεότητα σύμφωνα με, με το Βελιγράδι. Πολλά από τα προβλήματα της ασφάλειας θα παραμείνουν. Συμπεραίνω. Στο Κόσοβο ζούμε ένα πόλεμο συμβόλων. λιγότερο βίο από άλλες μορφές πολέμου. Παρ' όλα αυτά, πολύ συχνά φτάνει σε ένα επικίνδυνο κατόφλι και μπορεί να ξεσπάσουν βίες συγκρούσεις. Υπάρχει σημαντική απειλή από τους αλλοδαπούς μαχητές. Σημαντικό έβρος αποστεθεροποιητικών παραγόντων. Με τον κίνδυνο κάποια στιγμή η κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο. Χρειάζονται λοιπόν μηχανισμοί ασφαλείας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να ξεσπάσει η βία. Ο μετασχηματισμός του KSF είναι ένα σημαντικό θέμα. Μπορεί να είναι θεμητές οι φιλοδοξίες να γίνει πραγματικό στρατός, ο τρόπος όμως και ο χρόνος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα για να αποφευθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Η KFOR συμβάλλει σε ένα ασφαλές περιβάλλον και στην ελευθερία διακίνησης όλων των Κωσοβάρων, ανεξάρτητα από εθνότητα και ε, θρησκευμά. Και βεβαίως σημαντική είναι η Γιούλεξ ως δεύτερος που καλείται να απαντήσει στις ε, προκλήσεις ασφαλείας. Η Γιούλεξ, ξαναλέω, είναι ο δεύτερος security responder, παρεμβαίνει όταν αυξάνεται η πίεση στην ε, αστυνομία του Κόσοβου. Αν δεν ήταν, ε, αν δεν είναι μάλλον σε δυνατότητα η Γιούλεξ να αντιμετωπίσει, έρχεται η k σειρά της k Θα πρέπει να εκτιμηθούν και οι διώξεις που ασκεί το ειδικό δικαστήριο μέσα σε ένα ενδεχόμενο σενάριο για το μέλλον του Κωσόβου. Και κλείνω με μία εικόνα που βλέπετε αμερικανικό ελικόπτερο πίσω και ένα κροατικό ελικόπτερο μπροστά και ένα ελβετικό λίγο πιο πίσω. Άρα η K4 που χρησιμοποιεί όλα αυτά τα αεροσκάφη είναι μια πραγματική πολυεθνική δύναμη που ξεπερνά τα όρια του ΝΑΤΟ, είναι σε θέση να διεξαγάγει πολύπλοκες στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα συνήθεια όρια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φώτιγκα. Ευχαριστώ στρατηγέ. Θα δώσω τώρα τον ε, λόγο στην ε, μόνιμη εκπρόσωπο του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ που υπήρξε και διαπραγματεύτρια της ένταξης στο ΝΑΤΟ του Μαυροβουνίου. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Η παρουσίασή μου θα είναι κάπως διαφορετική, δεν θα είναι τόσο στατιωτική. Θα χρησιμοποιήσω και εγώ PowerPoint. Να σας δώσω μια εικόνα των όσων πέρασε το Μαυροβούνιο στην, όσον αφορά την ένταξη στο ΝΑΤΟ και μετά να θέσω και το πλαίσιο ασφαλείας για τη γενικότερη περιοχή και το Μαυροβούνιο. Θα ξέρετε ότι σαν χώρα που ανεξαρτητοποιήθηκε το 2006 η διαδικασία εντάξεως στο ΝΑΤΟ ευθύς εξ αρχής ήταν το κλειδί για μας, για την ασφάλειά μας. Και αμέσως μετά την εξαρτησία γίναμε μέλος της σύμπραξη για την ειρήνη και ξεκινήσαμε προγράμματα συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ. Δεν θα επισέθω σε πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τα τακτικά προγράμματα, αλλά τότε τα προγράμματα βασιζόταν σε αυτό που θεωρούσαμε αναγκαίο για μας και σύμφωνα με το δικό μας ευχολόγιο και το ΝΑΤΟ βοηθούσε στο βαθμό του δυνατού. Στην αρχή λοιπόν είναι, κάναμε, δεν είχαμε κληρονομήσει μεγάλο στρατό και έπρεπε να ξυγχρονιστούμε και να περάσουμε κομμουνιστική εποχή ούτε να μετακινηθούμε από την α, κομμουνιστική εποχή σε νέα εποχή, έπρεπε να ξεκινήσουμε από το μηδέν στον αμυντικό τομέα και στον τομέα της ασφαλείας και να θεσπίσουμε νομοθεσία και να κινηθούμε αργά προς την υλοποίηση και εφαρμογή της νομοθεσίας. Η ασφάλεια και άμυνα ήταν ένα τμήμα της διαδικασίας και μόνο. Το άλλο φορούσε πολιτικά κριτήρια και το κράτος δικαίου. Βρήκαμε τρόπους αντιμετωπίσεως της διαδικασίας. Έμοιαζε και με την ενταξιακή διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίσαμε φορείς σε κρατικό επίπεδο, κυβερνητικό και σε άλλα επίπεδα με άμεση εμπλοκή των βουλευτών. Η διαδικασία ήταν το πρώτο ίμιση, θα έλεγα, της διαδρομής προς το ΝΑΤΟ. Πραγματική δουλειά ξεκίνησε όταν μπήκαμε στο σχέδιο δράσης για το ΝΑΤΟ, το MAP, που ήταν η βασική φάση προετοιμασίας πολύ πιο σοβαρή η προσπάθεια εκεί, εστιασμένο πρόγραμμα, υλοποιήθηκε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Όχι σύμφωνα με τις δικές μας απόψεις, αλλά σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ κινηθήκαμε για τα αναγκαία. Είχαμε τέσσερις βασικούς τομείς στη διαδικασία. Πρώτος, ασφάλεια, μεταρρύθμιση τομέα ασφαλείας, στρατός και άλλες πτυχές αμυντικές και μυστικέ υπηρεσίε για τη συλλογή πληροφοριών ασφάλεια, κράτο δικαίου, λεπτομερέστερα τώρα από ό,τι πριν, και το πολιτικό πλαίσιο μετά. Για μας ήταν σημαντικός ο πολιτικός διάλογος με τον ΝΑΤΟ. Αλλά το πιο δύσκολο ήταν η υποστήριξη, η δημόσια υποστήριξη, η υποστήριξη του λαού για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Περάσαν πέντε κύκλους ΜΑΠ. Στην άμυνα τι κάναμε εξασφαλίσαμε ότι εφαρμόζουμε τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, ότι υπήρχε διαλειτουργικότητα του στρατού. Δημιουργήσαμε δυναμικό, εξυγχρονίσαμε το στρατό, συμμετείχαμε σε αποστολές με την Ευρωπαϊκή με τον ΝΑΤΟ, με τον ΟΗΕ. Στον τομέα ασφαλείας και συλλογής πληροφοριών θεσπίσαμε νομοθεσία και αργά σταδιακά μεταρρυθμίσαμε την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, το Φορέ Εθνικής Ασφαλείας και άλλους φορείς κράτος δικαίου. Αυτό συνδεόταν με αυτά που συνέβαιναν στο μέτωπο ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιαστήκαμε επί μεταρρυθμίσεων και ανεξαρτησίας δικαστικού κλάδου κατά πολέμη διαφθοράς και εγκλήματος και όλες τις στοιχείες που αφορούν την ενταξιακή μας πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρθώσαμε να αρμονίσαμε, εφόσον είμαστε μικρή χώρα κιόλα και δεν έχουμε τόσα πολλά, τόσο μεγάλο προσωπικό, εναρμονίσαμε λέγω αυτό που κάναμε στον τομέα με αυτά που κάναμε στην Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν κοινέ προσπάθειες, κοινό προσωπικό όσον αφορά το μέτωπο ΝΑΤΟ και το μέτωπο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποστήριξη του λαού ήταν το πιο δύσκολο. Ξεκινήσαμε με τον ατρίτο του πληθυσμού να μας υποστηρίζει να είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, πολιτικός πώς, αν μεταφραστεί στην άποψη των πολιτικών κομμάτων, υποστήριξαν διπλάσια. Ποιο ήταν το πρόβλημα, να δούμε γιατί συνέβαινε αυτό. Επίσης, πώς να εντοπίσουμε τα προβλήματα και τι να κάνουμε. Εντοπίσαμε τα προβλήματα. Κυρίως, ο κόσμος δεν είχε αρκετή ενημέρωση όσον αφορά το τι σήμαινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ, τι σημαίνει το ΝΑΤΟ, οι απόψεις βασιζόταν σε ψυχροπολεμική άποψη για τον ΝΑΤΟ και τον ρόλο που διαδραμάτισε. Ποτέ βέβαια δεν πρέπει να παραμελεί κανείς ε, και τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργήθηκαν την παρέμβαση των ΝΑΤΟ το 1999. Υπήρχε άγνοια, ελλειπής πληροφόρηση, ε, προκαταλήψεις έντονες κατά του ΝΑΤΟ αποστατική βάση που λέγανε ότι θα κατασκευάσουν βάσει σε τουριστικές περιοχές, θα καταστρέψουν ε, το περιβάλλον, ε, οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ θα απολαμβάνουν τιμωρησίες κλπ. Εντοπίσαμε τα προβλήματα, διαμορφώσαμε στρατηγική και είδαμε από την αρχή ότι δεν μπορεί να είναι κυβερνητικό το πρόγραμμα και το σχέδιο. η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ήταν κρατικός στόχος. Κινηθήκαμε σε κυβερνητικό επίπεδο αρχικά για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Συμμετείχαν πολιτικά κόμματα, βουλευτέ, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, πανεπιστημιακοί, ΜΜΕ και ΜΚΟ. Που έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με την κυβέρνηση. Και κάναμε τα πάντα για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σήμαιναν όλα αυτά σε δύο χρόνια από όταν εστιάσαμε τις προσπάθειες και στείλαμε σαφή μηνύματα, καταφέραμε να ανεβάσουμε την υποστήριξη σχεδόν στο 50%. Και η τάση ήταν ανωδική. Αυξήθηκε η κατανόηση. Θα προτιμούσαμε βέβαια να φτάναμε ακόμα ψηλότερα. Όμως αυτή ήταν η εμπειρία του Μαυροβουνίου και λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματά μας όσον αφορά τα συναισθήματα που είχε ο λαός και όχι μόνο ορθολογική προσέγγιση αυτό δεν ήταν καθόλου παράξενο αυτή η αντιμετώπιση και άλλες χώρες αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα τώρα εδώ και 10-15 μέρες είμαστε μέλη και όσο περνάει ο χρόνος που είμαστε μέλη αργά-αργά αυτές οι ιδέες και οι προκαταλήψεις θα διαλυθούν σχετικά με την ε, δισταγμούς και ανησυχίες για το να είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Είχαμε και θέματα νομικά να λύσουμε όσον αφορά το ΝΑΤΟ, παρόμοια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αλλά πολύ μικρότερο τομέα. έχει δικό του κεκτημένο το ΝΑΤΟ. Έπρεπε να εναρμονίσουμε το κεκτημένο του ΝΑΤΟ με το δικό μα εθνικό κεκτημένο. Μετά από αυτού του τέσσερους κύκλου MAP που περάσαμε, που ήταν ανοιχτή διαδικασία, και τα έγγραφα ήταν δημόσια, που δεν είναι εύκολο για περίπτωση, την περίπτωση του ΝΑΤΟ. Είχαμε τακτική υποβολή αναφορών και επικοινωνία με το αρχηγείο των ΝΑΤΟ για ενημέρωση. Μετά από αυτό είχαμε στον ΠΕΣ, είχαμε μια σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ και ένας νέος μηχανισμός αναπτύχθηκε εκεί. Ενδεδικοποίηση εστιασμένων συζητήσεων ήταν ο τίτλος. Εδόθηκε στο Μαυροβούνιο μια περίοδος ενός έτους να εστιαστούμε επί συγκεκριμένων τομέων. Τεσσάρων τομέων που έπρεπε να γίνουν προσπάθειε. Και κατά τη διάρκεια του έτου αυτού ήταν εντατικότατη η επικοινωνία με τον ΝΑΤΟ. Κάθε μήνα τουλάχιστον. Αναλύαμε διάφορες λεπτομέρειες για διάφορα ζητήματα που εκκρεμούσαν. Και αυτό που βοήθησε πολύ ήταν η ειλικρινέστατη και πολύ ανοιχτή προσέγγιση του ΝΑΤΟ και απαντήσεις μας έδινε το ΝΑΤΟ για το τι έπρεπε να κάνουμε. Όλα αυτά οδήγησαν μετά την περίοδο αυτή ότι το Μαυροβούνιο πληρούσε τα κριτήρια και το Δεκέμβριο του 2015 προσεκλήθημεν να γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ. Πολύ σύντομα μετά από αυτό και εδώ έπαιξε ε, είχε σημασία ο διαπραγματευτικό ρόλο που αναφέρθηκε, παρόλο που δεν μοιάζει με την ανταξιακή πορεία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεγράφει το πρωτόκολλο προσχώρηση μεταξύ Μαυροβουνίου και ΝΑΤΟ. Εκεί διαπραγματευτήκαμε το πώ θα λειτουργήσει το όλο ζήτημα. Μετά από αυτό, το Μαυροβούνιο ξεκίνησε τη συμμετοχή στι εργασίε του ΝΑΤΟ κατά 70% στι επίτροπέ, σε όλου του τομεί του ΝΑΤΟ, όχι στα πάντα, διότι υπάρχει διαφορά μεταξύ προετοιμασίας και πλήρους συμμετοχής, πλήρους μέλους. Όσο επικυρώνωνε το πρωτόκολλο προσχώρησης στα κράτη του ΝΑΤΟ, εμείς στις Βρυξέλλες στο αρχηγείο αρχίσαμε να μαθαίνουμε τη διαδικασία, να συμμετέχουμε σε όλα τα σώματα και φορείς, να παραλαμβάνουμε όλα τα έγγραφα και ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε και εδώ και στη χώρα μας, στα διάφορα υπουργεία, στους κυβερνητικούς θεσμούς να προετοιμαζόμαστε ούτω ώστε όταν έρθει η μέρα και γίνουμε πλήρη μέλη όλα να εκτυλιχθούν ομαλά. Και αυτό ήταν και πάλι δύσκολο για μια μικρή χώρα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα για μια μικρή χώρα, αλλά ήμασταν επιτυχέστατοι. Και όπως ξέρετε στις 5 Ιουνίου, από όταν, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία κύρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Μαυροβουνίου, εμείς επικυρώσαμε τη συνθήκη της Ουάσιγκτον, παρόμοιο έγγραφο με πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Και τότε γίναμε μέλος του ΝΑΤΟ στις 5 Ιουνίου. Εν γέννη λοιπόν, αυτή ήταν η μεταμορφωτική διαδικασία που αφορούσε κυρίως την κοινωνία μας και τους θεσμούς. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν σημαντικότατη και πήγαινε χέρι με χέρι διαδικασία με τη διαδικασία εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα συμπλήρωναν το ένα το άλλο και αποτελούσαν ένα τμήμα αργής πρόοδου, παρά τις διαφορές της δύο διαδικασίες βέβαια. Τώρα, πού βρισκόμαστε τώρα, πριν αναφερθώ στα θέματα ασφαλείας και στα ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Ήταν σαφέστατο ευθύς εξ αρχής και αυτό που κάνουμε τώρα είναι να λέμε ότι είναι ένα νέο κομμάτι της όλης προσπάθειας η συμμετοχή του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταρρυθμίσεις είναι σε σχέση με αυτό που απαιτείται για να είμαστε επιτυχές μέλος του ΝΑΤΟ. Ούτε οι μεταρρυθμίσεις για μας να γίνουν, να γίνουν στη χώρα μας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν την κοινωνία. Και αυτό περνάει και μέσα από τη διαδικασία την ενταξιακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το τι είναι σημαντικό και τι μεταρρυθμίσεις απαιτούνται ακόμα για τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, προσαρμόζεται ο στρατός μας, αυξάνει το δυναμικό του και είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί απλώς να σταματήσει να λήξει όταν γίνει μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Μίλησα για επικοινωνία δημόσια ανοιχτή, επικοινωνία με το κοινό, αυτή συνεχίζεται. Εξηγούμε τι σημαίνει το ότι είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, τι κάνει το ΝΑΤΟ και οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ στις οποίες συμμετέχουμε τώρα. Σε εθνικό επίπεδο, πολύ σημαντικό, είναι το θέμα και το, το κράτος δικαίου και προχωράμε εκεί και στα πλαίσια της διαδικασίας ενταξιακής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένταξη στο ΝΑΤΟ, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοήθησε πάρα πολύ, οδήγησε σε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Το κλειδί ήταν να κατανοηθεί ότι αυτό δεν γίνεται σαν αυτός σκοπό. Θέλαμε να αλλάξουμε εμεί η κοινωνία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ μας δίνουν απλώ κατευθυντήριες γραμμές. Και έχει καλά αποτελέσματα αν κάνεις εθνικό επίπεδο σωστή προσπάθεια. Και αυτό το διαβιβάσαμε στον κόσμο μέσω της διαδικασίας για την ένταξη του ΝΑΤΟ, εφόσον ολοκληρώθηκε και επιτυχώς. Δουλειά μας τώρα είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πλήρη επίγνωση των μελών και έχουμε επίγνωση των, συγγνώμη, επίγνωση των ευθυνών που έχουμε σαν μέλος του ΝΑΤΟ, να είμαστε ένα πολύ αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια, υπήρξαν στο δρόμο μας προς το ΝΑΤΟ, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα και σήμερα μπορούμε να πούμε θέλαμε να γίνουμε μέλος. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αποφάσισαν ότι η προθυμία μας, η δουλειά μας, η αφοσίωσή μας ήταν κάτι καλό και γι' αυτό γίναμε μέλος. Το μέλλον θα αποδείξει ότι δεν θα μετανιώσει καμία από τις δύο πλευρές. Τώρα τι σημαίνει το ότι είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια του Μαυροβουνίου σε περιφερειακό και ευρύτερο επίπεδο. Εξυπακούεται και για αυτό το βασικό λόγο ξεκινήσαμε τη διαδικασία σαν χώρα. Ξεπακούεται λέγω ότι θα βοηθήσει και θα παγιώσει τη σταθερότητά μας, την ασφάλειά μας και έμεσα συνεπάγεται ότι αυτό θα επηρεάσει και την οικονομική μας ανάπτυξη. Σίγουρα χρειάζονται και άλλες μεταρρυθμίσεις και δοθέντος του υφισταμένου ενθουσιασμού εν της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσουμε, ενθουσιασμού για να συνεχίσουμε μπορούμε να συνεχίσουμε. Διότι αποδείξαμε ότι όταν δουλεύει κανείς σοβαρά υπάρχει αποτέλεσμα. δουλειά, η σκληρή δουλειά αποδίδει. Τεράστια σημασία να είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Έχουμε μια θέση στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, έχουμε φωνή, συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων, μοιραζόμαστε πληροφορίες, προωθούμε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή και όπως ακούσατε υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα στην περιοχή Υπάρχουν πολλά προβλήματα και πέρα από την περιοχή. Πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, προβλήματα ε, κυβερνοαπειλών, απειλών στον κυβερνοχώρο, κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια χώρα ή από μια περιφέρεια. Ε, βοηθάει η Ένωση και γι' αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Επίσης η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ σημαίνει πολλά για την περιοχή. Όπως και όταν μπήκε η Κροατία και η Σλοβενία είχε σημασία και η Αλβανία αργότερα ε, μετά το Μαύρο Όσο εντα, ε, εντασσόμεθα σαν χώρε στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλύτερο για την περιοχή. Αυτό είναι αυταπόδεικτο, ε, είναι αυτονόητο για, ότι είναι σημαντικό η σταθερότητα στην περιοχή. Δεν θα επιληθούν προβλήματα ασφαλείας στην περιοχή, βοηθάει όμως. Το ότι είμαστε μέλος είναι ένα καλό παράδειγμα και δείχνει ότι είναι αξιόπιστη η ενταξιακή προοπτική και αυτό είναι σημαντικό για τις χώρες της περιοχής. Τώρα, όσον αφορά περιφερειακή ασφάλεια, δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τα περισσότερα στοιχεία ήδη έχουν αναφερθεί. Ανεξάρτητα από την πρόοδο που υφίσταται, υπάρχουν προβλήματα που αναφέρθηκαν. Κάποια προβλήματα συγκεκριμένα για κάποιες χώρες, κάποια αντιμετωπίζονται από όλες τις χώρες. Το Μαυροβούνιο πιστεύει ότι ο καλύτερος μοναδικός τρόπος πέρα από το να κάνουν τη δουλειά τους και τους αριθμίσει στις χώρες είναι να υπάρχει σαφής προοπτική για τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες. Και δεν πιστεύω μόνο αυτό, αλλά χρειάζεται σαφής επαφή με τις δύο οργανώσεις, τους δύο οργανισμούς αυτούς σε πρακτικό επίπεδο και πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει επαφή με τις χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ μπορούν να συνεργαστούν. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία σε όλα αυτά. Είναι ξεχωριστοί οργανισμοί με διαφορετικές διαδικασίες αλλά με κοινές αξίες πολλές από αυτές. Και όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια παρόμοιες απόψεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικοδομητικό. Βοηθάει. Η ασφάλεια στην περιοχή είναι κάτι αλληλένδετο. Τα προβλήματα ξεχυλίζουν από χώρα σε χώρα. Δεν θα αφεληθεί καμία χώρα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια άλλη. Κανείς από εμά δεν είναι πάντα ασφαλής ή σταθερός όταν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αν δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αν όλη η περιοχή δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρέσβυρα και να αρχίσουμε τώρα την συζήτηση με τον κύριο Στέτινα, αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, περιμένω λίγο να φορέσουν τα ακουστικά οι συνάδελφοι. Με ενδιαφέρει κυρίως η παρέμβαση του κυρίου Φούγκο. Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο που επιτυγχάνει ε, η K-Force το Κόσοβο. Θέλετε να επαναλάβω αυτό που είπα. Κύριε Κωνστάτηγε, εκφράζω την εκτίμησή μου. Α, ίσως υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Με ακούτε τώρα. Συνεχίζω στην ε, μετρική μου γλώσσα. Έχω μία ερώτηση για τον ε, κύριο Φουνγκό. Πριν όμως ε, σας θέσω την ερώτηση, στρατηγέ μου, επιθυμώ να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ε, μακρότατη αυτή αποστολή της K4 που είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής. Μιλήσατε για πόλεμο συμβόλων, για ε, σύγκρουση συμβόλων και σύγκρουση οραμάτων για το Κόσοβο. Υπενθυμίζω σε όλους ότι όχι και τόσο, στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν η Επιτροπή μας είχε προτείνει τον κύριο Χαβιέρ Σολάνα, πρώην Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον είχαμε συναντήσει μάλλον, και ένα από τα θέματα που είχαμε συζητήσει τότε ήταν τι γινόταν τότε όταν αποφάσισε ο Σολάνα να στείλει βομβαρδιστικά στην Ιουκοσλαβία. Εγώ κατενόησα ότι τα δύο οράματα, η θετική αξιολόγηση της απόφασης εκείνης για τον βομβαρδισμό της ε, πρώην Ιουκοσλαβίας και το αρνητικό αρνητική άποψη εξακολουθούν να είναι ζωντανές και οι δύο αυτές απόψεις, θέσεις, οράματα εξακολουθούν να είναι ζωντανές. Γνωρίζω ότι στη χώρα μου, την τσεχική δημοκρατία, το παράδειγμα του βομβαρδισμού της ε, δημοκρατίας χρησιμοποιείται ακόμη ως όπλο κατά όλων εκείνων που λένε όχι στο ΝΑΤΟ και όχι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Βαν Όρντεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τους στρατηγούς και την πρέσβη. Δεν θα απογοητεύσω τους συναδέλφους και θα εκφράσω τις επιφυλάξεις που έχω για την ΚΕΠΑ. Ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει ε, να κατανοήσουμε την πραγματικότητα που δεν ε, ε, τα παρουσιάζει όλα υπό άριστο φως. Στον τομέα που συζητάμε σήμερα το πρωί, η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ικανότητες άμυνας σε, έχετε σε μια περίπλοκη κατάσταση. Βλέπω την επιχείρηση Άλθια, παραδείγματο χάρη. Έχουμε τουλάχιστον πέντε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεισφέρουν στην επιχείρηση Άλθια. Στην αποστολή ε, K4 εκεί κοντά πάλι που είναι επιχείρηση του ΝΑΤΟ περιλαμβάνονται ε, τέσσερις ε, ουδέτεροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε τους λόγους γιατί έχουμε χωριστή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και Ιδίω τώρα που το Μαυροβούνιο είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι θα είχε νόημα να έχουμε ένα συντονιστικό κεντρικό σημείο για τις επιχειρήσεις σε αυτή την περιφέρεια. Και το μεγάλο πλεονέκτημα για τον αναπληρωτή, είπα, το συμμαχικό διοικητή του ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη ε, είναι το ότι ε, μπορείτε με το ρόλο αυτό να προωθήσετε μια τέτοια τάση. Υπάρχουν και ε, τα δύο θέματα τα οποία παραμένουν σε ερωτήματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Στατηγέ, ποια θεωρείτε τα βασικά ζητήματα της στρατιωτικής παρέμβασης. Ε, τα στρατεύματα δεν ε, συμμετέχουν σε μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ε, παίζουν το ρόλο, έχουν αποτρεπτικό ρόλο. θα μπορούσε να υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της άρσης των ναρκών. Έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό εδώ ε, επί πολλά χρόνια και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζουμε μετά από 20 χρόνια να συζητάμε για ένα πρόβλημα με νάρκε στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Θυμάμαι πριν από χρόνια θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ένοπλε δυνάμεις της Βοσνίας τουλάχιστον, αν δεν έκαναν τίποτα άλλο, τουλάχιστον θα ξεκαθάριζαν τι νάρκες. Και τώρα 20 χρόνια αργότερα ακόμη δεν το έχουν κάνει τι μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πολλά χρόνια, για, πολλά χρήματα συγγνώμη, για τέτοιες δράσεις άρσης ναρκών. Τέλος, ξέρω ότι δεν είναι απολύτως της αρμοδιότητά σας, αλλά σκεφτόμαστε και το θέμα των μελλοντικών σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προσβλέπουμε σε μια θετική εταιρική σχέση μετά τον Brexit. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς μία σχέση με την, ευρωπαϊκή, με την στρατιωτική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία χρήσιμη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα εντό παρενθέσεως χωρίς ε, να πολυενθαρρύνουμε τέτοιες τάσεις, αλλά αν έχετε κάτι να σχολιάσετε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος, ο κ. Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ όλους τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας για τις παρεμβάσεις τους και έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον προς τον στρατηγό Εβερντ για την Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευτυχώς η χώρα σιγά σιγά Ε, γίνεται μια χώρα που όχι μόνο καταναλώνει υπηρεσίες ασφάλειας, αλλά και η ίδια παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας. Η ερώτησή μου είναι πώς ε, αξιολογείται τη λειτουργία, την απόδοση των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας και Ζεγοβίνης ε, δέκα χρόνια μετά την ενοποίησή τους. Δεύτερον, αν θέλετε να σχολιάσετε θα την αποκαλούσα αντιφατική συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης τον ε, Ιανουάριο όταν έγινε ο διαχωρισμός με την Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Και τρίτον, πιστεύετε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, θα επεκτείνει την εντολή της Eurofor και τι επιχειρήματα έχετε για την ε, επέκταση αυτή. Προς τον υποστάτηγο Φούγκο θα ήθελα να πω ότι ε, είχα επισκεφθεί το Κωσυφοπέδιο και ε, πάντοτε με εκπλήσει ε, πολύ ευχάριστα η δραστηριότητά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δράση σας και παρακαλούμε συνεχίστε το εξαιρετικό σας έργο. Προς την κυρία Πρέσβη θα ήθελα να πω ότι ε, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για συγχαρητήρια προς το Μοντενέγκρο για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολλά θέματα και ένα βασικό μήνυμα πιστεύω. Δηλαδή, ο λαός της χώρας αποφασίζει για τη μελλοντική εξέλιξη της χώρας και όχι κάποιος άλλος απ' έξω, όσο και να προσπαθούν ε, οι απ' έξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα μελλοντικά υποψήφια κράτη για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ακόμη και αν δεν είχατε παρουσίαση PowerPoint, η παρουσίαση σας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κούκανο, κύριο Φρόιν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι αντάξιος των ε, προηγουμένων ομιλητών. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά πριν περάσω στην ερώτησή μου, θέλω να μιλήσω για κάτι που είπε ο κύριος Βαν Όρντεν. για την απομάκρυνση των αρκών στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Ως δημοσιογράφος, πριν από 10 χρόνια, όχι 20 χρόνια που είπατε εσείς, κάλυψα αυτά τα θέματα και ε, έχω πολύ ζωντανές μνήμες όταν παρακολουθούσα σε ένα ναρκοπαίδιο κοντά στο Σεράγεβο τη διαδικασία που επρόκειτο να γίνει για την άρση των ναρκών και με εκπλήσει και εμένα όπως και εσάς ότι ε, το θέμα αυτό παραμένει ανεπίλητο μετά από 20 χρόνια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι είναι απολύτως απαράδεκτο το ότι δεν έχει επιληθεί το θέμα αυτό. Ε, περνώ τώρα στο άλλο μου θέμα. Υπήρξε ένα θέμα όσον αφορά τη συμμετοχή της Αυστρίας στην K4 και εγώ είμαι Αυστριακός Ευρωβουλευτής και γι' αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δική σας αντίδραση. Όπως ξέρετε, η Τουρκία μπλοκάρει το πρόγραμμα στρατιωτικης συνεργασία Αυστρία Αυστρίας-ΝΑΤΟ, το οποίο μπορεί να επηρεάζει τα αυστριακά στρατεύματα της ΚΕΙΦΟΡ στην περιοχή και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα. διότι η Τουρκία δεν θέλει να συμμετέχει η Αυστρία σε αυτή την περιοχή. Είναι σημαντική η συνεισφορά της Αυστρίας στην ΚΕΙΦΟΡ. Δεν έχω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία αυτή τη στιγμή. 300, 400 στρατιώτες ή κάτι τέτοιο. Σχετικά σημαντική λοιπόν η συμμετοχή μας. Και αφού μιλήσατε για τις προκλήσεις για την K4 ε, στο προσεχές μέλλον, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το θεωρείτε και αυτό μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσετε μέσα στους προσεχείς μήνες. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια λύση για το αδιέξοδο αυτό μεταξύ Τουρκίας και ΝΑΤΟ ή μήπως είναι μεταξύ Τουρκίας και Αυστρίας ή Τουρκίας, Αυστρίας και ΝΑΤΟ. Θα ήθελα κάποιο σχόλιο για το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και την κυρία Πρέσβη και τους δύο στρατηγούς για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση που μας έκαναν. Ε, θα είμαι σύντομος. Θα απευθύνω μία ερώτηση στον Στρατηγό Everard υπό την ε, ιδιότητά του ως ε, D-Secure για το εάν και κατά πόσον το ΝΑΤΟ εκτιμά αυτή τη στιγμή ότι και για την Βοσνία Ερζεγοβίνη αλλά και για το Κωσυφοπαίδιο υπάρχει εξωτερική στρατιωτική απειλή. Επίσης ήθελα να ρωτήσω την κυρία Πρέσβη το εξής. Ποια σκοπιμότητα ασφαλείας θέλει να ικανοποιήσει η χώρα σα με την ένταξή τη στο ΝΑΤΟ. Είπατε προηγουμένω κι εσεί ότι ο συνασπισμό εκείνο ο οποίο ε, επετέθη στη χώρα σα ήταν το ΝΑΤΟ. Τι άλλαξε αυτή τη στιγμή και η χώρα σα θέλει να διασωθεί από ποια απειλή γενομένη μέλο του ΝΑΤΟ και από την άλλη πλευρά υποχρεώνοντα το ΝΑΤΟ αν χρειαστεί να ενεργοποιήσει και το άρθρο 5 περί συλλογική ε, ασφάλειας κατά αυτής της απειλής που απειλεί τη χώρα σας. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Μποστινάρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις. Και οι τρεις για τον ε, κύριο Έβεραλτ. Πρώτο, ρωσική στρατιωτική παρουσία είναι μόνο περιορισμένοι, είναι κόγχοι ή είναι ε, κάποια άλλη που βρίσκεται ας πούμε σε αγωγό, έρχεται. Δεύτερον, η ειναι καποιοι αλλοι που βρισκεται ας πουμε σε αγωγο ερχεται δευτερο η ευρωπαικη ενωση θα πρέπει να ζητήσει από όλε τι υποψήφιε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων να ευθυγραμμίσουν τι εξωτερικέ πολιτικέ του με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια από τα πιο πρώτα ή δυνατόν βήματα για να αντιμετωπιστούν κενά ή προβλήματα. Γιατί υπάρχουν χώρες και φωνές από την περιοχή που λένε ναι, ναι, να το κάνουμε, αλλά κάποια άλλη φάση. Αυτή η αμφισημία σε περιόδους αβεβαιότητας είναι σημαντικό πρόβλημα. Τέλος, τι θα πρέπει να κάνουν οι χώρες των Βαλκανίων για να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια της περιοχής με εφαρμογή μορφών στρατιωτικής συνεργασίας. Θυμούμε παλαιότερα αρχές δεκαετία του 90, ή μάλλον τέλη δεκαετία του 90, αρχέ των 2000, να υπάρχουν πολλά σχέδια συνεργασία μεταξύ των στρατών των, ε, της περιοχής αυτής και των αμυντικών τους τομέων. Σήμερα υπάρχει σημαντικός βαθμό εμπιστοσύνη ανάμεσα στα στρατιωτικούς τους ο κύριος Ζαϊρανόπουλος. Απευθύνομαι στους δύο στρατηγούς του ΝΑΤΟ με δύο πολύ μικρές ιστορίες. Το 1999, όταν τα ανατοϊκά στρατεύματα περνούσαν για το Κόσοβο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκη, ο ελληνικός λαός με επικεφαλή κομμουνιστές αντιστάθηκε και έστειλε τα ανατοϊκά στρατεύματα στην τουριστική Χαλκιδική. Πριν από τρει εβδομάδες, στα πλαίσια μια άσκηση του ΝΑΤΟ, στρατιωτικά αγήματα του ΝΑΤΟ κινήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα και έξω από την Κοζάνη 100 κομμουνιστέ ανάγκασαν ένα στρατιωτικό αγήμα του ΝΑΤΟ με όπιστε να φύγει. Το επόμενο Σάββατο, και κλείνω με αυτό, στρέψτε τα μάτια στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδε εργαζόμενοι και συνδικάτα, επειδή το ΝΑΤΟ συνεχίζει να ματοκυλάει τα Βαλκάνια, χιλιάδε εργαζόμενοι και συνδικάτα θα σα στείλουν το εξή μήνυμα. Η Ελλάδα έχει πολύ ωραίες παραλίες και θάλασσες. Ενημερώστε τους στρατιώτες να πάρουν και μαγιό μαζί τους, γιατί εκεί θα είναι η κατάληξή τους. Εκεί θα είναι ο προορισμός τους. Σε χλωρό κλαρί, ο ελληνικός λόγος κομμουνιστές δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. That the list. Ευχαριστώ. Εδώ κλείνει ο κατάλογος ε, των ε, ομιλητών. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα ε, στους πανελίστ με την ίδια σειρά πρώτος ο κ. Σέβρατ, μετά ο υποστάτηγος κ. Φούγκο και μετά η κυρία Πρέσβης. Ευχαριστώ. Μακρά λίστα ερωτήσεων. Αν δεν απαντήσω πλήρως, σας παρακαλώ ε, υπενθυμίστε μου. Σε ό,τι αφορά την απειλή και τη στρατιωτική εμπλοκή στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Μου φαίνεται πιθανό να αναπτύξουμε δυνάμεις εάν αντιληφθούμε ότι επιδεινώνεται η πολιτική κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσία τάξη. Αυτά έχουν αποτέλεσμα ε, στην εμπιστοσύνη. Σε ό,τι αφορά τις χερσαίες νάρκες, δικαίως ανησυχούμε. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Αφενός είναι η ποσότητα ναρκών που έχουν ε, ναρκοθετηθεί. Αλλά και το δεύτερο είναι και το πού ακριβώς έχουν γίνει ναρκοθετήσεις. Υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία από ναρκοθέτησης γύρω από διάφορους μη κρατικούς και από την κυβέρνηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, την οποία εμείς στηρίζουμε. Χρειάζεται μια νέα όθηση και στην αναθεώρηση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ζητήσει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ρωτήσατε για τον μελλοντικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενδεχόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είμαι Βρετανός αξιωματικός, αλλά έχω και η ιδιότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την 35η μου σταδιοδρομία στο Βρετανικό στρατό, που νομίζω ωστόσο ότι αποτέλεσε και θαυμάσια προετοιμασία για το ρόλο που έχω αναλάβει ως αναπληρωτή ΣΑΚΕΡ. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στην κοινή αμυντική προσπάθεια θα πρέπει να συνεχίσει. Για παράδειγμα, όπως σε περιοχές όπως η Balkan Reserve έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε δυνάμεις ταχύτατα και θα πρέπει να τη διατηρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την Βοσνία Ζεγοβίνη που πέρασε από το να καταναλώνει υπηρεσίε ασφάλεια στο να παρέχει υπηρεσίε ασφάλεια, αυτό συμβαίνει σε έναν αριθμό επιχειρήσεων και αυτές, αυτοί οι σχηματισμοί που αναπτύσσονται λαμβάνονται από τις τρει εθνοτικές κοινότητες και δίνουν, δείχνουν σημαντική ε, δέσμευση και στράτευση. Τους επισκέφθηκα την ε, δύναμη της Βοσνίας του στο Αφγανιστάν πρόσφατα. Ασφαλώς και αντιμετωπίζουν τοπικές πιέσεις που τους δυσχεραίνουν τη ζωή, αλλά πάλι εκεί η λύση είναι περισσότερο ε, μεγαλύτερη πολιτική ενότητα η εντολή των Ηνωμένων Εθνών και γιατί θα πρέπει να τα ανανεώσουμε. Ελπίζω, εάν κοιτάξετε το χρονοδιάγραμμα, να αντιληφθείτε ότι η στρατηγική αναθεωρή, strategic review, όταν θα ξανασυζητηθεί σε φόρουμ όπως το δικό σας, δεν θα είναι πριν από τις αρχές του 2018. Και θα είναι πλέον σαφές αν επιθυμούν να ανανεώσουν την εντολή τα Ηνωμένα Έθνη. Εφόσον επανεξετάζεται η εντολή, αυτό θα πρέπει να γίνει σε, με συζητήσεις σε βάθος, χωρίς την αφαίρεση επιλογών. Η συμμετοχή της Αυστρίας. Αυτό είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Εγώ θα σημειώσω μόνο ότι Τούρκοι και Αυστριακοί συνεργάζονται θαυμάσια μέσα στα πλαίσια της δυναμιάς μας, του ΝΑΤΟ δηλαδή. Ελπίζω ότι θα υπερισχύσει ο ρεαλισμός και θα ληφθεί η ορθή απόφαση στην πολιτική, στο πολιτικό επίπεδο. Οι απειλές μέρος του σχεδιασμού μας στρέφεται γύρω από την ασφάλεια και την αποτροπή. Ρωσική στρατιωτική παρουσία, κάποιος με ρώτησε. Δεν με εκπλήσει ούτε και με ανησυχεί η ρωσική εμπλοκή στην περιοχή των Βαλκανίων, διότι έχουν ε, μακρά ιστορική παράδοση. Στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει διαφορετική, διαφορετικός τρόπος. Μέσω διαλόγου πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μεγαλύτερη συνεργασία και αλληλοκατανόηση με τη Ρωσία. Το άλλο για την ευθυγράμμιση νομίζω είναι ζήτημα περισσότερο για την κυρία Μογκερίνη. Τέλος, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Το μέγα θέμα που προκύπτει μέσα από τη Security Review είναι οι δραστηριότητες που διεξάγονται και όπου δεν γνωρίζει ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται διμερώς ασφαλώς και είναι μια σημαντική χειρονομία αλληλεγγύης με την χώρα αυτή. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τον συντονισμό όλων των προσπαθειών μας για την Βοσνία Ζεγοβίνη και νομίζω ότι πρόκειται για πραγματική αναγνώριση ότι το μέλλον εξαρτάται από την συνεργασία με εταίρους και σε ολόκληρο τον πλανήτη. στη βάση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό αυτό. Τέλος, α, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής έφυγε τώρα. Εγώ ήμουν στο Κόσοβο το 1999 και θυμούμαι ότι οι Έλληνες 90% ήταν αντίθετοι με την συμμετοχή της K4. Και όμως συμμετέσχουν με ένα τάγμα και τελικώς η αποδοχή ήταν της τάξης του 90%. Αποδοχή πλέον 90%. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ε, πιο σύντομος ο κατάλογος, είμαι τυχερός. Να σας πω ότι είναι το μεγαλύτερο στράτευμα το αυστριακό από ε, τις χώρες και δεν υπάρχουν ε, αμφισβητήσεις όσον αφορά την ε, αποτελεσματικότητα των δυνάμεων κάτω από μένα είναι ε, αυστριακός στρατηγός και καθοδηγεί τουρκικές μονάδες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την εκτέλεση των διαταγών και την εκτέλεση των αποστολών. Στον κύριο Στετίνα, ο πόλεμος των συμβόλων δεν σχετίζεται με τον βομβαρδισμό, είναι η επιδέξη εκμετάλλευση μικρών γεγονότων ή συμβόλων που είναι διάσπαρτα στο κοσυφοπέδιο για να αυξηθεί αντιπαράθεση σε ρητορικό επίπεδο. Ποιο είναι το θετικό. Όλοι οι παρόντες φορείς στο κοσυφοπέδιο, οι διεθνείς βοηθούν να διατηρηθεί η αντιπαράθεση σε ρητορικό επίπεδο. Αυξάνεται το επίπεδο επιλύσεως των προβλημάτων θα πρέπει να δρά η διεθνής κοινότητα άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων. you, Ευχαριστώ, Στρατηγέ. Κυρία Πρέσβυρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ έχω λίγες ερωτήσεις να απαντήσω. Θα είμαι σύντομη λοιπόν. Ποιες είναι οι απειλές που βλέπουμε ως μέλος του ΝΑΤΟ και αν υπάρχει και κάποια απειλή που βλέπει το άρθρο 5. Οπότε δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί. Οι απειλές ε, βάσει του άρθρου 5 είναι σοβαρές απειλές ε, που μπορεί να περιλαμβάνουν στρατιωτικούς ή εδαφικούς κινδύνους και ε, είναι μια κατάσταση που δεν νομίζω ότι είναι πιθανή ούτε ε, όταν δεν ήμασταν μέλο του ΝΑΤΟ, ούτε ως ε, μέλη του ΝΑΤΟ. Και περνώ και στο δεύτερο τμήμα της ερώτησης, ε, ποιοι είναι οι στόχοι μα ω προς την ασφάλεια ως μέλη του ΝΑΤΟ. Μα ακριβώ αυτό, ότι δεν είναι πλέον... Δεν υπάρχει πλέον μια τέτοια πιθανότητα γιατί έχουμε ζήσει τον πόλεμο στα Βαλκάνια και η ιδιότητά μας του μέλους του ΝΑΤΟ Μα εγγυάται ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Η στερεωτική απειλή δεν είναι η μόνη απειλή. Υπάρχουν πολλές απειλές τρομοκρατίας, ε, κυβερνοπολέμου. Δεν είναι άσπρο-μαύρο αυτή η κατάσταση. Όλες οι χώρες είτε μέλο του ΝΑΤΟ, είτε μη μέλο του ΝΑΤΟ, είτε στα Δυτικά Βαλκάνια, είτε εκτό Βαλκανίων. όλε οι χώρε είναι εκτεθειμένε σε τέτοιου κινδύνου. Αλλά για να είμαστε όσο δυνατόν καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου κίνδυνου, ακόμη και για τι μεγαλύτερε χώρε, αλλά ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια μικρή χώρα, το να είναι κανεί μέλο ε, μια αμυντική συμμαχία όταν έχει την τεχνογνωσία, όταν έχει τη βοήθεια, όταν μαθαίνει πώ να επαυξάνει το ίδιο δυναμικό της ε, έχει πολλά ωφέλη. Δεν είναι ότι περιμένουμε από το ΝΑΤΟ να μας σώσει από απειλές, αλλά θέλουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας ως μέλος του ΝΑΤΟ μαζί με τους συμμάχους μας για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να αμυνθούμε έναντι ιεσδήποτε απειλής. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι δεν υφίσταται κάποιο κίνδυνο υπό την έννοια του άρθρου 5 για την περιφέρεια, αν και ποτέ κανεί δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις καταληκτικές μας παρατηρήσεις και θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Κούζο Περμόη, εκ μέρους της ΑΦΕΤ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής, όλους τους περιορισκομένους για τα σχόλιά σας. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις όταν συζητάμε την κατάσταση ασφαλείας στα Δυτικά Βαλκάνια. και τις σχέσεις των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να παρέχουμε υποστήριξη στις χώρες αυτές. Η περιφερειακή συνεργασία είναι σημαντική και αποτελεί τη βάση για την ε, ε, διαρκή σταθερότητα στην περιφέρεια. Είναι σημαντικά λοιπόν όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα για το έργο το οποίο αναμένεται από εμά στο μέλλον. Ευχαριστώ και ξαναδίνω το λόγο στη Συμπρόεδρο κυρία Φώτιγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου τη Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ήθελα και εγώ, Υποεπιτροπή Συγγνώμη Ασφάλεια και Άμυνα, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω του διακεκριμένου συμμετέχοντε να, τα συγχαρητήριά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας, ε, στρατηγέ Everard ε, και υποστρατηγέ Φούγκο. Και θα ήθελα και προς την ε, κυρία Πρέσβη να πω ότι και εγώ προέρχομαι από μια πρώην κομμουνιστική χώρα και συμφωνώ απολύτως με τη διαδικασία μετασχηματισμού της χώρας σας. και με την προσπάθειά σας να προσεγγίζετε όλο και περισσότερο τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Κλείνουμε λοιπόν την πρωινή μας ε, συνεδρίαση με αυτά τα σχόλια και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το απόγευμα Έχουμε επίσης ενδιαφέροντα σημεία στην ημερήσια διάταξη, μια, την παρουσίαση μιας μελέτης για την αντιτρομοκρατική συνεργασία με τις χώρες της νότιας γειτονίας. Θα γίνει και ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο King που θα μας ενημερώσει για ό,τι νεότερο υπάρχει για την Ένωση Ασφάλειας. Και έχουμε και άλλα σημεία ίσονος σημασίας δεδομένων ε, των δύο πρώτων σημείων που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και αύριο το πρωί έχουμε επίσης ε, συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την ε, Επιτροπή Άφετ που ήταν μαζί μας και τους προσκεκλημένους μας.